Okay, everybody, could you take your seats, please? Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, εντάξει, μπορώ να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασης. Έχουμε πρώτα την έγκριση της διάταξης. Αντιρρήσεις, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Σημείο 2, ανακοινώσεις της Προέδρου. Τίποτα δεν έχω να σας πω και με μεγάλη χαρά σας το λέω. Πάμε λοιπόν στο σημείο 3, η ανταλλαγή απόψεων με το Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, τον κύριο Άγχελ Γκουρία. Είναι η πρώτη φορά, κατά τη θητεία αυτή τουλάχιστον, που ένας εκπρόσωπος του ΟΣΑ έχει έρθει σε συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Αυτό μας την μεγάλη χαρά. Έχουμε κάθε διάθεση για καλύτερη συνεργασία. Φυσικά έχουμε διαφορετικά θέματα τα οποία μας απασχολούν στη Μέση Διάταξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΩΣΑ θα κάνει μια παρέμβαση περίπου 15 λεπτών <clears throat> και μετά, όπως γίνεται συνήθως, ως ήθιστε θα έχουμε ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων και αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των βουλευτών που θα θέσουν ερωτήματα. Ενδεχομένως θα σας ομαδοποιήσω για να δώσει μια απάντηση ο κύριος Γκούρια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ, χαιρόμαστε που, πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Έχουμε, είχαμε μια πολύ καλή σχέση με τον κύριο Πέτερινγκ, με τον κύριο Μπούζεκ και τον κύριο Σούλτς που θα δω αύριο και με την πρόεδρο την κυρία Sharon Bowles που συναντήσαμε μαζί με τους πρόεδρους όλων των επιτροπών και επειδή έχουμε τα ίδια θέματα που μας απασχολούν, την ίδια μέρημνα, πολλές φορές τους ίδιους στόχους, βέβαια δεν είμαστε πάντα εισακουστοί από το ΕΚΟΦΗΝ. Έχω τον Άντωνη Γκούρτς εδώ, ο οποίος είναι επικεφαλής της, ε, των δημοσίων σχέσεων και, των, και της επικοινωνίας στον ΩΣΑ. Η κυρία Γκαμπρία Λαράμος είναι σέρπα για τους G20, επίσης είναι μαζί μας. Ο Σεμπαστιαν Μπάρνς επίσης ο οποίο είναι εμπειρογνώμων για τα οικονομικά θέματα. Ξέρουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι δικοί σας εκπρόσωποι στον ΩΣΑ. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να χαιρετήσουμε την παρουσία τους. Μεγάλη η χαρά μου λοιπόν που μπορώ να λάβω το λόγο ενώπιον της Οικονομικής και Νομισματική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω το λόγο ενώπιόν σα, βέβαια. Αλλά αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι ένα πιο έντονο διάλογο ο οποίο θα οδηγήσει σε μελλοντικέ ανταλλαγές απόψεων. Για μα είναι κρίσιμη σημασία, ζωτική σημασία η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 21 από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του όσα όπως γνωρίζετε. Από τα 34 λοιπόν μέλη του ΟΣΑ, 21 ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η σχέση μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κέρυας σημασίας. Είναι η πιο σημαντική κοινοβουλευτική συνέλευση λοιπόν που έχουμε να αντιμετωπίσουμε λόγω του μεγάλου αριθμού μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΩΣΑ αλλά και λόγω των αρμοδιοτήτων που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την ε, νομοθετική διαδικασία και με την κανονιστική διαδικασία που έχει στον οικονομικό στίβο. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην ιστορία μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύση σε τεράστιες οικονομικές προκλήσεις και προκλήσεις απασχόλησης. Όλα αυτά μέσα σε μια προσπάθεια να βρούμε λύσεις, να δώσουμε ελπίδα στους πολίτες και να διατηρήσουμε τη δημοκρατική μας νομιμοποίηση. Δεν έχει τελειώσει φυσικά η κρίση ακόμα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακόμα βραχυπρόθεσμες προκλήσεις. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα λιγάκι πρόσφατα. Υπήρξε μια λύση προσωρινή για το θέμα της Ελλάδος που έχει καταπραίνει λιγάκι τις αγορές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει την απαραίτητη ρευστότητα για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου μισό τρισεκατομμύριο. Η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και αρχίζουν να φυτρώνουν και πάλι μπουμπούκια από την άλλη άκρη του Ατλαντικού βέβαια. Αυτό το περιμέναμε να γίνει πριν από τρία χρόνια, γίνεται αυτή τη στιγμή. Όλος ο κύκλος λοιπόν έχει καθυστερήσει λιγάκι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν τελειώσει όλα αυτά τα προβλήματα. Παραμένει το θέμα της εμπιστοσύνης στην αγορά που είναι περιορισμένη και κυρίως δεν έχουμε πολύ καλές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη στο παγκόσμιο στερέωμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πηγή της κρίσης, να ξεπεράσουμε τις οικονομικές και δημοσιονομικές ανισότητες μέσα στην παγκόσμια οικονομία, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του υπορβελικού χρέους, να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και δημιούργησης θέσεων απασχόλησης που είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το δημόσιο χρέος είναι κάτι που δεν το έχουμε επιτύχει πλήρως ακόμα. Προσβλέπουμε στη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ στα, επόμενε επόμενες και ένα τείχος ανάσχεσης είναι απαραίτητο να γίνει ακόμα πιο στεναρό για να προστατευτούμε έναντι των αγορών. Χρειαζόμαστε, όπως θα έλεγε κάποιος, την μητέρα όλων των τείχων ανάσχεσης για να μπορέσουμε να δώσουμε και τη δύναμη πυρός στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Όσο πιο ισχυρό το τείχος ανάσχεσης λοιπόν, τόσο πιο απίθανο θα είναι ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε μια μελλοντική κρίση. Όσο πιο εύκαμπτα λοιπόν είναι τα συστήματά μας, τόσο πιο εύκολα θα προσπαθήσουν να προσπαθήσουν ορισμένοι να δοκιμάσουν το στοίχημα. Παρά το γεγονός ότι η κρίση στην Ευρώπη είναι το κύριο μέλημά μας, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε άλλες παγκόσμιες πραγματικότητες. Μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξαν εξελίξεις στις αναδυόμενες οικονομίε οικονομίες του κόσμου, οι οποίες μετατόψαν το ε, κέντρο βάρου βάρους της παγκόσμιας οικονομίας προς τα νότια και τα ανατολικά. Οι αναδυόμενες οικονομίες πέρασαν από το 36% το 1961 όταν δημιουργήθηκε ο ΩΣΑ στο 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ, και παρά το γεγονό ότι οι δυνατότητε οικονομική ανάπτυξη για τι αναδυόμενε αυτέ χώρε συνδέεται με τι δικέ μα προοπτικέ, το δυναμικό ανάπτυξή του ξεπερνάει το δικό μα. Έχουμε λοιπόν μια τάση ανάπτυξη η οποία είναι πολύ ισχυρότερη για τι χώρε αυτέ. 1,5% είναι η μεσοπρόθεσμη προβλεπόμενη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,5% το χρόνο. Ενώ οι χώρε αυτέ αν συγκρούμε και με τις ΗΠΑ που βρίσκονται στο 2%, οι αναδυόμενες χώρες έχουν ένα δυναμικό ανάπτυξης που μπορεί να φτάσει το 8% και το 9% στην περίπτωση της Κίνας. Μετατοπίζεται λοιπόν γεωγραφικά ο πλούτος από 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2,5% ίσως στις ΗΠΑ, αλλά 8 με 9% στις αναδυόμενες χώρες. Πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη στις χώρες αυτές τέσσερις φορές παραπάνω από τις παραδοσιακές ε, βιομηχανικές χώρες. Όταν η Ευρώπη θέλει να έχει τους καλύτερους εγκεφάλους, τα μεγαλύτερα προσόντα, αντιμετωπίζει ανταγωνισμό όχι μόνο από την Αμερική και την Καναδά, αλλά και από την Ινδία και την Κίνα. Οι φοιτητέ της Κίνας και της Ινδίας είναι όλο και καλύτεροι από τους Ευρωπαίους. και στις κατατάξεις τα πανεπιστήμια οι φοιτητές των πανεπιστημίων από τις αναδυόμενες χώρες ξεπερνούν την Ευρώπη αν εξαιρέσουμε τις σκανδιναβικές χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται στο επίπεδο των χωρών αυτών σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, τη συμμετοχή στο ενεργασιακό χώρο. Μειώνονται οι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χαμηλότερο επίπεδο από τι ΗΠΑ και την Ιαπωνία ή την Κορέα. Για να φέρουμε μια χώρα που δεν είναι από τις πιο ανεπτυγμένες στον κόσμο. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν σημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα, ένα σκόδον κινδύνου για την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί περισσότερο για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι όπως αυτά που ένιωσε η Αμερική όταν εκτοξεύτηκε ο Σπούτνικ από την Ρωσία το 1957 και τότε ξεκίνησε το σχέδιο για να, στείλει, να στείλουν οι έναν άνθρωπο στο φεγγάρι μέσα στην επόμενη δεκαετία. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν υψηλή ανταγωνιστικότητα, υψηλή παραγωγικότητα για την Ευρώπη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό και να αντιμετωπίσει και κοινωνικές προκλήσεις. Γιατί δεν έχουμε μονάχα χαμηλή ε, οικονομική μεγέθυνση, αλλά και αυξανόμενη ανισότητα. 24 άτομα, εκατομμύρια άτομα είναι άνεργα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενεργεία των νέων ξεπερνάει το 20% και φτάνει και μέχρι και το 50% σε ορισμένε χώρε. Επειδή είναι πιο δύσκολο βέβαια να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης όταν υπάρχει λιτότη σε επίπεδο δημοσιονομικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη χρειάζεται μια ατζέντα για ανταγωνιστικότητα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί σε αυτή την παγκόσμια πρόκληση σε σχέση με τον χώρο της απασχόλησης. Αυτό σημαίνει πρέπει να προχωρήσουμε σε διαφορετικέ αλλαγές, να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη συμμετοχή στο χώρο της εργασίας, περισσότερη ελευθερία στην παροχή υπηρεσιών. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σύστημα των ε, συντάξεων, να αυξήσουμε τα προσόντα, να βοηθήσουμε την καινοτομία και το επιχειρήμα. Και το μεγάλο πρόβλημα με τα διαρθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κυρία Μπάους, είναι ότι πράγματι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δέσμοι. Ως αντιμετωπίζουμε με μονομένα μέτρα για την αντιμετώπιση αλλαγών στις διαθρώσεις, αυτά δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο ως δέσμοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα αυξηθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε και ένα στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίο θα συμβάλλει σε αυτή την ανάπτυξη. Οι φιλόδοξε μεταρρυθμίσει στο διαθετικό επίπεδο δεν είναι μονάχα για να φέρουν μια ανάκαμψη σε μια δύσκολη εποχή, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τι ακαμψίες οι οποίε δημιούργησαν τι ανισότητε, οι οποίε έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα, ώστε να είμαστε και καλύτερα προετοιμασμένοι για μελλοντικού κλειδονισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πραγματικό σύμφωνο ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό ο ΩΣΑ είναι έτοιμος να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία όχι μόνο των ευρωπαϊκών μελών του, αλλά και των άλλων χωρών του κόσμου που μπορούν να συγκριθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι πηγή έμπνευση. Όταν εργαζόμαστε με την Ισπανία και την Ιταλία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν θα πρέπει να συμβάλλουν σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και όχι μόνο η Ιταλία και η Ισπανία. Να φέρω την προσοχή σας σε μία περίπτωση που βεβαίως ε, ε, στην περίπτωση της Ισπανίας έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες σε σχέση με την ε, ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά ήταν μία από τις, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ακόμα δεν, έχουν, δεν, έχει, δεν έχει γίνει σωστή εκμετάλλευση και πλήρης εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα οι απαιτήσει ε, τη υφιστάμενη ενιαία αγορά θα πρέπει με αποτελεσματικότερο τρόπο να εφαρμοστούν. Δεύτερον, η Ευρώπη χρειάζεται ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο σχετικά με την διασυνοριακή οικονομία. Και τρίτον, χρειάζεται μεγαλύτερη πρόοδος ε, όσον αφορά ε, ειδικέ διατάξεις για συγκεκριμένους τομείς όπως ας πούμε διασυνοριακές προμήθειες και διαγωνισμοί, αύξηση οικοδόμηση ικανοτήτων κτλ. Μονάχα 3% ε, των πολιτών της Ευρώπης που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας δουλεύουν σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωση ενώ στην, στον ίδιο ε, τομέα πληθυσμού έχουμε 5% ε, μετανάστευση από τρίτες χώρες. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε και οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις να έχουν έχουν την δυνατότητα να βρουν το σωστό ε, προσωπικό. Γιατί ξέρετε φτάνουμε σε αυτό το παράδοξο. Πολύ συχνά ε, λέμε μα δεν έχουμε εσωτερικό δυναμικό έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στι ανάγκε μα. Πρέπει να το εισάγουμε. Επίσης, ε, ε, σαν απόρρια αυτής της κατάστασης ε, προκύπτουν περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλη ανάπτυξη και άλλες οι οποίες υπολείπονται. Θα πρέπει επίσης να δούμε από πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εστιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια στοιχεία όπως είναι ας πούμε η, τροπο, αλλαγή του τρόπου συνταξιοδότησης κτλ. Επίσης θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στους εργαζόμενους ε, να βρεθούν αντιμέτωποι με την ε, παγκοσμιοποιημένη ε, οικονομία έτσι ώστε να μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Μέχρι τώρα η, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τη δυνατότητα να ελκύει ταλέντα και εγκεφάλους. Αυτή τη στιγμή δεν, είναι... δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Επίσης η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη κατάρτισης σε δεξιοτήτων κτλ. θα πρέπει να ε, αυξηθεί θα πρέπει οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν τώρα τα θεμέλια έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η βάση για την καλή ε, ανάπτυξη. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, οι καινοτομίες, θα πρέπει να υπάρχουν οι δεξιότητες, οι απαραίτητες έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να προχωρήσει. Επίσης θα πρέπει να αρθούν όλα αυτά τα διαρθρωτικά εμπόδια τα οποία ακόμα αποτελούν πρόσκομα στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Τρίτον, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το εργασιακό δυναμικό, ε, να δοθεί μεγαλύτερη βάση στην κατάρτιση, την εκπαίδευση και την χρησιμοποίηση τη σωστή των ικανοτήτων ε, του ε, εργασιακού δυναμικού. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσεχτεί ιδιαίτερα ε, η γύρανση του πληθυσμού με όλες τις εκφάνσεις αλλά και όλες τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει ε, και τις οικονομικές βεβαίως επιπτώσεις που μπορεί η γύρανση αυτή να έχει. Ε, πρέπει να πω ότι αυτή η γύρανση και οι επιπτώσεις της ε, αφορούν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρτογραφήσει καλύτερα το θεσμικό και εργασιακό πεδίο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες, τις τεράστιες προκλήσεις που έχει απέναντί της. Ο Winston Churchill είπε ότι οι ε, απεσιόδοξοι βλέπουν δυσκολίες σε κάθε ευκαιρία, ενώ οι αισιόδοξοι βλέπουν ευκαιρίες ε, σε κάθε δυσκολία. Ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και να σας πω ότι ο οργανισμός που εκπροσωπώ είναι πάντα στο πλευρό σας και ευελπιστεί σε καλύτερη και στενότερη συνεργασία στο μέλλον. Και λόγω του ίδιου του λειτουργήματος του οργανισμού και λόγω ε, της ίδιας της ουσίας του ε, είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τα μέλη μας, άρα και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπα και στην αρχή, τα περισσότερα μέλη μας είναι ταυτόχρονα και μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξουν στο μέλλον καλύτερες πολιτικές για καλύτερη ζωή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μα πάντα ο καφέ σε άκυρη στιγμή έρχεται. Τέλος πάντων. Έτσι είναι η ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίσατε την τελευταία μας συνάντηση που ήταν νομίζω ένα άτυπο εκοφήν. Όταν νομίζω πάλι αγώνα δύναμε για την επίλυση της κρίσης και το κεφάλαιο των τραπεζών, τύχη προστασίας κτλ. Πάλι τα ίδια θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και τουλάχιστον τα πράγματα έχουν πάει εκεί όπου προσπαθήσαμε να τα κατευθύνουμε πριν από αρκετό καιρό. Λοιπόν, έχω αρκετού στο κατάλογο των, στον κατάλογο των ομιλητών, οπότε παρακαλώ να είστε σύντομοι πρώτα απ' όλα για το ΕΛΚ. Παύλο, σας ευχαριστώ Σάρον. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, παρουσία σας, αλλά και για τις εξαντλητικές ε, ε, επεξηγήσεις τις οποίες αναφέρατε. Είπατε ότι υπάρχουν διαστάσεις ανάμεσα στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της, του ΟΣΑ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτές ε, οι διαστάσεις, αυτές οι διαφορές φαίνεται ότι μεγαλώνουν τον τελευταίο καιρό. Σε τι οφείλεται αυτό. Ενώ υποτίθεται ότι ε, η αξιοπιστία βεβαίως ε, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Να σας πω απλώς ότι καμιά φορά αυτό σχετίζεται με τη στιγμή στην οποία εκδίδουμε τις προβολές αυτές και όταν βγάζουμε τα μοντέλα μας κτλ. Η μεγαλύτερη ανησυχία μου δεν είναι ε, οπωσδήποτε η τυχόν διαφορά, αλλά ότι μετά από αυτή την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση εξακολουθούμε να θεωρούμε πως ε, εργαζόμαστε χωριστά. Ε, εγώ θεωρώ πως η κρίση συνέβη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνής ε, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ε, ILO, τα κτλ. δεν ε, συνεργάζονταν αρκετά. Ο καθένα ήταν στο γραφείο του και εργάζονταν στο πλαίσιο της εντολής του και κανείς δεν είδε το τρένο που ερχόταν. Και θα ήθελα να πω πως κάτι στο οποίο επιμένουμε στις ετήσιες ε, συναντήσεις μας με την Αγγέλα Μέρκελ και με τους G20 που μιλάμε για το ζήτημα αυτό της σύγκλησης ή συνεργασίας. Αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε πως συμφωνούμε. Και πρέπει να πω πως ε, αυτό οπωσδήποτε είναι αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο και προκαλεί σκέψη. Γιατί ξαναγκάζει τον κόσμο να σκεφτεί, μα γιατί υπάρχουν αυτέ οι διαφορέ. Κάποιε σχετίζονται με τι υποθέσει που κάνουμε, κάποια μοντέλα είναι βραχυπρόθεσμα, άλλα μακροπρόθεσμα, άλλε προβολέ, ε, άλλε είναι προσωμιώσει, ε, άλλε είναι εξηγήσει του τι έχει μόλι συμβεί. Δεν βλέπω να έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές. Αλλά να σας πω κάτι άλλο και με αυτό θα τελειώσω τους τελευταίους μήνες. Το επίπεδο επιδίνωσης των προβλέψεων, όλο χαμηλότερα, χαμηλότερα, χαμηλότερα, τι γινόταν. Δευτέρα ε, είχαμε κάτι χαμηλότερο και Παρασκευή είχε αναθεωρηθεί και αυτό προς τα κάτω. Εάν δείτε δηλαδή ένα διάστημα τριών μηνών μεταξύ της τελευταίας προβολής ε, του Δουνουτού και της ε, τελευταίας του ΟΣΑ ή αντιστρόφως ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όσο πιο πρόσφατη τόσο και χειρότερη. Κυνηγούσαμε την ουρά μας. Τώρα θα έλεγα πως θα γίνει λίγο το αντίθετο. Σε κάποιες περιπτώσεις ειδικά όσον αφορά τη ΣΥΠΑ που είναι κάπως καλύτερα θα δούμε κάποια βελτίωση. Αλλά τα βασικά στοιχεία δεν είναι τόσο σαφή σήμερα. Γι' αυτό θα ε, κοιτάμε στοιχεία ανάκαμψης χωρίς να είμαστε πεπισμένοι πως έχουμε μια γενικευμένη τέτοια κατάσταση. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικό ακόμα. Εγώ προτιμώ ακόμα να είμαι επιφυλακτικό αντί να πω πως ξεπεράσαμε την κρίση. Δεν ξεπεράσαμε την κρίση όταν έχουμε κατά μέσο όρο 10% ανεργία που αυξάνεται στην Ευρώπη, 20% μέσο όρο ανεργία των νέων, 30-40% σε κάποιες χώρες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει ε, την κρίση. Οπότε για να μην είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι ή κάποια σημάδια να το θεωρήσουμε πως είναι η αρχή της ανάκαμψης, ε, δεν θα το έκανα εγώ. Εγώ θα έλεγα να είμαστε καλύτερα επιφυλακτικοί. Σας ευχαριστούμε για τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της ε, συναδέλφου Φερέιρα που ήθελε να σας θέσει το ερώτημα αυτό. Αναφερθήκατε σε μια στιγμή σπούτνικ για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη φτάνει στο 1,5%. Αλλά βλέποντας τα συστατικά στοιχεία αυτής της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον βιομηχανικέ ε, ε, βιομηχανικές επενδύσεις με σημαντικό η απόδοση. Επίσης ε, ε, στον ιδιωτικό τομέα γενικά οι επενδύσεις είναι πολύ μικρές και ότι στον δημόσιο τομέα οι περικοπές είναι πάρα πολύ μεγάλες λόγω της κατάστασης. Όσον αφορά τώρα τους φορείς ανάπτυξης ε, έχουμε την εντύπωση ότι μάλλον με, τις, με τα νέα μέτρα θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις των καταναλωτικών συνηθιών. Επομένως δεν νομίζω Νομίζουμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για μεγάλη και, θε, και έτσι, θεαματική ανάκαμψη. Ερώτηση λοιπόν. Είναι λογικό να ε, συνεχίζουμε να μην θέλουμε ε, τέτοια ε, πολιτική προϋπολογισμού. Εμείς πρέπει να σας πω ότι είμαστε σαν σοσιαλδημοκράτες πολύ ορθολογικοί και πιστεύουμε ότι στους ε, λειτουργικούς προϋπολογισμούς θα πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Ε, επομένως, πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να πάρουμε αντικυκλικά μέτρα όσον αφορά τις επενδύσεις, κυρίως δεν τις δημόσιες επενδύσεις και εν τη αυτή περιπτώση ποια είναι η άποψή σας σχετικά με, το, με την πρόταση που κάνουμε, δηλαδή ε, να αφαιρεθεί από, τους, από τις ε, επενδύσεις το ποσοστό επενδύσεων ε, για την ε, ανάπτυξη έτσι ώστε να μπορέσουν μέσω των προϋπολογισμών τους τα κράτη να προετοιμάσουν το μέλλον. Ε, the question... Το ερώτημα του γιατί λέτε πως οι επενδύσεις ε, δεν σχετίζονται πλέον και δεν αντιδρούν στα επιτόκια. Θεωρώ πως δεν αντιδρούν στα επιτόκια γιατί τα ζητήματα τα σχετικά με την επενδυτική απόφαση είναι πολύ σοβαρότερα από τα επιτόκια. Και είναι ακριβώς το επίπεδο αβεβαιότητας που είναι τόσο ψηλό και το επίπεδο δυσπιστίας ή το επίπεδο εμπιστοσύνη αν θέλετε είναι τόσο χαμηλό. Αυτή η κρίση είναι και κρίση εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα, στα κόμματα, στα κοινοβούλια, Στι κυβερνήσει σε όλα αυτά που έχουμε οικοδομήσει τόσα χρόνια. Γι' αυτό είναι τόσο σοβαρή. Και αυτό είναι τόσο ανησυχητικό. Και γι' αυτό ακριβώς ε, έχει την δυνατότητα να προξενήσει τόσο πολύ ζημιά. Και έχει ήδη προξενήσει. Γιατί δεν έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα ακριβώς της εμπιστοσύνης αυτής. Τώρα, να περάσω κατευθείαν στο ε, ουσιαστικό ερώτημά σας που λέτε πως ε, λόγω όλων αυτών των πραγμάτων και επειδή βλέπουμε πως ε, είναι της μόδας ε, η λιτότητα και όλα αυτά τα πράγματα που είναι στα πρωτοσέλιδα. Όχι, δεν συμφωνώ πως μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρος τις επενδύσεις και θα το θεωρήσουμε κάτι ξεχωριστό από τον γενικό προπολογισμό. Όχι, όλα πρέπει να είναι στον προπολογισμό γιατί η πηγή χρηματοδότησης είναι ίδια. Ξέρουμε πως οι επενδύσεις είναι κάτι καλό και στο μέλλον θα φέρουν ανάπτυξη, αλλά εντωμεταξύ πρέπει να χρηματοδοτηθούν και πρέπει να πάει κανείς στην αγορά. Και ιδεοδός, μέσω μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία θα χρηματοδοτήσουν. αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα πως οι κυβερνήσεις εξοδεύουν περισσότερα. Ε, το να το ε, πούμε και να το τονίσουμε αυτό θα μας οδηγήσει σε μια και να το, να το αγνοήσουμε συγχωρείτε θα μας οδηγήσει σε μια έκρηξη την οποία θα έχουμε προετοιμάσει οι ίδιοι. Μπορούμε να το διαχωρίσουμε αλλά είναι νομίζω απολύτως θεμητό να εξηγήσουμε και να διαχωρίσουμε τους διαφορετικούς τύπους δαπανών που πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Και επίσης ε, κάμια φορά είναι οριακή η κατάσταση. Δηλαδή κάποιες δαπάνες ε, στην εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθούν ε, τρέχουσες δαπάνες, αλλά κατά βάση θα πούμε πως οτιδήποτε σχετίζεται με έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση κτλ. είναι μια επένδυση για το μέλλον. Αλλά είναι δύσκολο να φανταστούμε πως ε, δεν θα επενδύσουμε στον ότι δεν θα μπουν, δεν θα ενταχθούν ε, οι επενδύσεις στον προπολογισμό. Ή θα λέμε πως είναι μόνο υλικά, κτίρια, μηχανήματα και όλα αυτά με ένα μαγικό τρόπο θα βρεθούν εκτός προπολογισμού. Δεν μπαίνει η υγεία στον προπολογισμό, γιατί είναι μεγάλη επένδυση. Ναι, είναι επένδυση στο σημαντικότερο πράγμα που υπάρχει στους ανθρώπους. Τι ε, πιο σημαντικό υπάρχει. Αλλά μετά λέμε να, να το αφήσουμε και αυτό κατά μέρο, Δεν μετράει και αυτό στον προπολογισμό. ω έλλειμμα. Ε, μα οι επενδύσει στην υγεία και στην ε, εκπαίδευση τυχαίνει να είναι οι μεγαλύτερε μαύρε τρύπε που έχουμε σε κάθε χώρα όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά. Οπότε, εάν αποφασίσουμε να ε, κάνουμε, να χτίσουμε μόνο δρόμους ή βιολογικούς καθαρισμούς, Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά εγώ θεωρώ πως πρέπει να μπαίνουν όλα σωστές, να έχουμε σωστές ε, μεθόδους υπερπολογισμού, να υπάρχει διαφάνεια, μην προσπαθείτε να κρύψετε τίποτα από τον καταναλωτή, να εξοδεύετε σωστά τα χρήματά τους, του φορολογούμενου, και να υπάρχει διαφάνεια. Και επίσης επειδή πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Και γιατί ειλικρινά. Μπορεί κανένα ε, να δώσει το δικό του ορισμό για να είναι πιο άνετα, αλλά ε, για, αυτού αυτούς που το προσπάθησαν στο παρελθόν και σας διαβεβαιώ πως κάποιοι το προσπάθησαν, κάποια μέρα ξύπνησαν και ανακάλυψαν πως ε, η κατάσταση ήταν εφιαλτική. Και αρκούσε λίγες από αυτές τις επενδύσεις να μην ε, αποδώσουν και να έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια οικονομικά. Δεν νομίζω πως είναι αυτό το πρόβλημα δηλαδή να τα διαχωρίσουμε. Δεν κερδίζουμε τίποτα και θα είναι ε, αντικατοπτρισμός, μια οφθαλμαπάτη. Μάλιστα όλοι ξυπνάνε τώρα και θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, οπότε θα σας ακούσουμε δύο-δύο. Βολφ Κλίντς και Φιλίπ Λαμπέρτς, οι επόμενοι δύο. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι για το ότι ήρθατε εδώ σήμερα και ελπίζω να είναι αυτή η αρχή τακτικών ε, συναντήσεων. Αναφέρατε ήδη... Ε, με ακούτε? Ωραία. Αναφέρατε ήδη το βασικό θέμα της ερώτησής μου, δηλαδή έχουμε μια βασική κρίση εμπιστοσύνης και έχω την εντύπωση πως ε, ο τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης δεν βελτιώνει την κατάσταση αλλά την επιδεινώνει κάνουμε συνεχώς προτάσεις και λαμβάνουμε αποφάσεις οι οποίες μετά από λίγο είναι πάλι ξεπερασμένες. Και είπατε στις αρχικές σας παρατηρήσεις πως θα πρέπει αυτό ακριβώς το τείχος προστασίας να επεκταθεί για να μας παίρνουν σοβαρά οι αγορές, τότε εγώ μπορώ να σας πω δεν θα τα καταφέρουμε. Έχουμε 503 εκατομμύρια, μετά θα πάει στα 750, μετά θα πάει στο τετράκι εκατομμύριο. Και μετά θα λένε 1,5 οι αγορές. Και μόνο κύκλους θα κάνουμε. Ο μοναδικός τρόπος να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη είναι να κάνουμε στα σοβαρά αυτό το οποίο θέλουμε. Δηλαδή λέμε θέλουμε να νοικοκυρεύσουμε τους λογαριασμούς, λέμε πως θέλουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, θέλουμε να λάβουμε μέτρα για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη κτλ. Αλλά δεν το κάνουμε. Δηλαδή, αν δείτε τη στιγμή που ε, δεν έχει στεγνώσει ακόμα το μελάνι στην υπογραφή του Πρωθυπουργού του κυρίου Ραχώη και ταυτόχρονα δηλώνει πως δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει, μα δεν δημιουργείται έτσι εμπιστοσύνη. Ε, και άκουσα από τους σοσιαλιστές πως ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε την ε, ανάπτυξη μέσω χρηματοδότηση. Μπορούμε πρώτα απ' όλα να προσπαθήσουμε χωρίς να ξοδέψουμε νέα λεφτά, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να υπάρξει μια πραγματικά ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες χωρίς να ξοδέψουμε τίποτα και παρόλα αυτά έτσι θα κινητοποιήσουμε την ανάπτυξη. Αλλά τι κάνουμε, αφήνουμε τα πάντα όσο έχουν. Δεν αλλάζει τίποτα. Και τέλο. Αναφερθήκατε στις απειλές, ε, στις ε, προκλήσεις που μας απειλούν από χώρες όπως η Κίνα, η Καναδάς και τα λοιπά. Συμφωνώ, ναι, αλλά εγώ επί μακρόν ε, ήμουν στον επιχειρηματικό βίο και πάντα είχαμε ως υπόδειγμα την Ιαπωνία μας έλεγαν πως είναι το μεγάλο υπόδειγμα και η μεγάλη απειλή και αν δεν κάναμε το χύψη θα μας ξεπερνούσαν οι Ιαπωνέζοι. Ε, νομίζω πως ε, αρκετά καλά τα πήγαμε στον ανταγωνισμό με την Ιαπωνία και δεν φοβάμαι και τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Απλά πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα οποία δηλώνουμε. Και τότε τα έχουμε καταφέρει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε. Καλώς ήρθατε κύριε Γκούρια στι Βρυξέλλε. Αγγλικά θα μιλήσω. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω ιδιαίτερα εδώ, γιατί ο ΙΣΑ... Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Είναι πάντα ο που φέρνει τις δυσάρεστες αλήθειες τους τελευταίους μήνες. Και η έκθεσή σας για την ανερχόμενη ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκθεσή σας επίσης για το γεγονός ότι έχουμε λησμονήσει τις προκλήσεις για το περιβάλλον και επίσης το γεγονός ότι πιέζεται πάντα για καλύτερη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα και θέλω να αναφέρω αυτό το οποίο έχετε ζητήσει να υπάρξει ένα όριο στη μόχλευση, όλα αυτά τα υποστηρίζουμε. Λέτε ότι είναι η στιγμή του Σπούτνικ για την Ευρώπη. Όχι μονάχα για τα θέματα ανάπτυξης, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης. Η δική μου ανάγνωση αυτής της ρίσης σας είναι σαν να λέτε ότι η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά για τη ρύθμιση στον τραπεζικό τομέα, για την αντιμετώπιση της καταστροφής του περιβάλλοντος για την εξάλληψη των ανισοτήτων. Είναι υπερβολικά αυτά που σας λέω ή αυτό ακριβώς λέτε κι εσείς. Όχι, όχι, δεν είσαστε υπερβολικός. Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά. Δεν είναι ότι δεν έχετε κάνει μονάχα πολλά. Είναι ότι όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Αυξάνεται η ανισότητα. Και πριν από την κρίση αυξάνονται οι ανισότητες έχουμε αυτό το έγγραφο που λέει είμαστε διχασμένοι, είμαστε σε διχόνοια και αυτό το, αυτή η δημοσίευση εξηγούσε γιατί αυξάνεται η ανισότητα στις ε, χώρες μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η σχέση εισοδήματος μεταξύ του χαμηλότερου 10% και του ανώτερου 10% είναι 7 φορές, 1 προς 7. Καλό ή κακό είναι αυτό. Δεν ξέρουμε. Στο παρελθόν όμως αυτό, το, αυτή η σχέση ήταν 1 προς 5, όχι 1 προς 7. Για τις καλύτερες περιπτώσεις είναι 7, ο μέσος όρος είναι 9, 1 προς 9, 1 προς 10, Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Τουρκία που φτάνει 1 από 14, στη χώρα μου στο Μεξικό 1 από 25, στην Βραζιλία είναι 50, μπορείτε να πείτε ναι, πολύ καλά τα καταφέρνουμε. Αλλά η τάση ίδια δεν είναι πολύ θετική. Αυξάνει παντού οι ανισότητες. Οι ανισότητες. Τον, η πιθανότητα να είναι κανείς φτωχός ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει το να μην είναι κανείς σε θέση να έχει βασικές υπηρεσίες, να μην έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες γίνεται όλο και πιο πιθανό για το περιβάλλον. Έχετε δίκιο. Έχουμε μόλις δημοσίευσει μια μελέτη πριν από λίγες μέρες που λέγεται «Οι συνέπειες της αδράνειας». Και το συμπέρασμά μας είναι πάρα πολύ απλό. Οποιαδήποτε δράση με τα σημερινά δεδομένα θα είναι πολύ πιο φτηνή για την ανθρωπότητα, θα κοστίσει λιγότερο στην ανθρωπότητα από ότι η αδράνεια. Αυτό που γίνεται στον τομέα της κλιματικής αλλαγής είναι ότι πάμε για μετοπική σύγκρουση με την φύση. Γιατί θα ξεπεράσουμε τα 450 ε, της εκατομμυρίης διοξίδιο του άνθρακος, αυτό θα αυξήσει, θα αυξήσει τη θερμοκρασία του πλανήτη και μετά, ακόμα και αν μειώσουμε την, ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, όσο καθυστερούμε περισσότερο, τόσο πιο πολυδάπανο θα είναι να επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα και το πιο πολύ θα κοστίσει. Οπότε οι στόχοι του 2050 μπορεί να μην έχουν κανένα νόημα απολύτω. και αυτό θα είναι μια μεγάλη απώλεια για την ανθρωπότητα. Η Ευρώπη τώρα πήγε πολύ καλά. Έδωσε το σωστό, τη σωστή κατεύθυνση για το σύστημα εμπορία εκπομπών, αλλά πρέπει να επανέλθουμε και να το υπογραμμίσουμε αυτό. Και για τι ανισότητες, οικονομικέ ανισότητε, έπραξε διάφορα πράγματα, αλλά αυτό θεωρείται ως μια παρακατιανή πολιτική, μια πολιτική που είναι δευτερεύουσα. Λέμε, εντάξει, αντιμετωπίστε την ε, οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και οι ανισότητες θα μειωθούν. Όχι, οι ανισότητες είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτόνομα τώρα πια. Για τον τομέα της ρύθμισης των τραπεζών, ιδίω για αυτόν τον τομέα θα έλεγα. Υπάρχει ένας αριθμός εθνικών ρυθμιστών μαζί με ένα μηχανισμό συντονισμού, αλλά το θέμα της επανακεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών δεν έχει κλείσει ακόμα και τα όρια στη μόχλευση τουλάχιστον χρησιμοποιήστε ένα συγκεκριμένο όρο. Μην βασίζεστε σε σταθμισμένα σε σχέση με το κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού, κάτι το οποίο είναι μια ασαφής έννοια τελικά. Χρησιμοποιήστε σαφή κριτήρια. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι δεν κάνετε αρκετά στην Ευρώπη. Να το πω αλλιώ. Μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα. Γιατί η ευρωπαϊκή οικοδόμηση είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το θαυμάσιο. Είμαι μεγάλος φαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θαυμάζω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1968 υπήρχε το ευρώ, το EQ, το, η Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα όταν κανείς δεν είχε σκεφτεί να εκδώσει ευρώ. Και στο Μεξικό τότε, εκείνη την εποχή το 1968, εκδίδαμε σε IQ ομόλογα. Ήμουν 18 χρονών τότε. Και εμείς βέβαια βρισκόμαστε στο Παρίσι, σε μια μεγάλη πόλη. Και να περάσω τώρα στο θέμα αυτό το οποίο για το θέμα της κρίσης εμπιστοσύνης. Το τείχος ανάσχεσης, όχι, δεν είναι κάτι το οποίο έχει καθυστέρηση, απλώς δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει το τείχος ανάσχεσης πριν από ένα χρόνο και δεν υπάρχει. Ίσως θα το φτιάξετε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ωραία, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το μέγεθος αυτού του τείχους ανάσχεσης. 500 δισεκατομμύρια. Κάποιος είπε ότι είναι 500 δισεκατομμύρια. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για 440, <clears throat> αλλά δεν είναι ζεστά και έτοιμα τα λεφτά αυτά, δεν είναι διαθέσιμα ακόμα. Η νέα διευκόλυνση η οποία προβλέπεται με αυτά που έχουν μείνει από, την παλαιά, από το παλαιό μέσο ή κάποια, μαζί με κάποια χρηματοδότηση από το Δουνουτού. Εντάξει. Δεν είναι ότι θα πούνε οι άνθρωποι έχουμε τώρα ένα τρισεκατομμύριο και αύριο θα έχουμε να κάνουμε τρία δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να δούμε ποια ομόλογα, ποια δάνεια θα οριμάσουν και θα φτάσουν στην εκπνοή τους τα επόμενα χρόνια. Αν θέλετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε τις αγορές, πρέπει να τους πείτε εδώ πέρα παίζετε με τα παιδιά μου. Και αν παίξετε με τα παιδιά μου, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Εάν θέλετε λοιπόν να κερδοσκοπείτε στα ομόλογα, να καταλάβετε ότι θα μειωθούν κάποια στιγμή οι αποδόσεις των ομολόγων και εσείς θα χάσετε τα λεφτά σου. Μα δεν κάνουμε λοιπόν αρκετά. Δεν χρησιμοποιούμε αρκετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χρηματοδοτεί, αλλά δεν χρησιμοποιεί τη δυνατότητα ομολόγων, αγορά ομολόγων στην αγορά. Ξέρω ότι αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Να σα πω όμω και το εξή. Ο κύριο Ραχώη που έλεγα προηγουμένω, αναφέρα, αναφέρατε κάποιε ανησυχίε για τον κύριο Ραχώη. Εγώ ήμουν μαζί μου. Δύο μέρε μετά που ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> και δώσαμε μια συνέντευξη τύπου και ήταν τότε ο υπέρμαχο τη προσαρμογή. Είπε ότι θα καταφέρω αυτό που μου έχουν πει, αλλά έχω κληρονομήσει 2,5% παραπάνω ε, χρέος σε σχέση με ΑΕΠ από ό,τι νόμιζα. Αλλά θα τα καταφέρω. Απλώς θα χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερο χρόνο, θα χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερη ευκαμψία τον πρώτο χρόνο, γιατί δεν μπορώ να απορροφήσω αυτά τα 2,5% μέσα σε ένα χρόνο. Εγώ υποστήριξα λοιπόν αυτή την προσέγγιση και θέλω να σας πω ότι από την πλευρά του κυρίου Ραχώη, του κυρίου Κίντος και των ηθινόντων στην Ισπανία, η εντύπωσή μου είναι ότι είναι όλοι τους προσιλωμένοι στο να μπορέσουν να επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους και θα το καταφέρουν γιατί τελικά τι είναι, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Όχι επειδή τους πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είχε ένα ρόπαλο πάνω το κεφάλι τους, όχι. Είναι γιατί κατανοούν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούν κρίση εμπιστοσύνης. Τέλος, είπατε ότι παλιά φοβόμασταν την Ιαπωνία. Αλλά η Ιαπωνία δεν τα κατάφερε καλύτερα από την Ευρώπη, όχι επειδή η Ευρώπη τα πήγε τόσο καλά, αλλά επειδή η Ιαπωνία έκανε λάθη. Μέχρι στιγμής όμως η Κίνα ακολουθεί μια πολύ αποφασιστική οδό έχουν πολλά προβλήματα σε εσωτερικό επίπεδο, πολλές εσωτερικές αντιφάσεις, αλλά δεν πρέπει να βασιζόσαστε στο ότι θα κάνουν λάθη. Αντιμετωπίστε εσείς τις δικές σας προκλήσεις και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Τώρα χρόνος πιέζει, οπότε θα ακούσουμε όλες μαζί τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Έχουμε 10 λεπτά και πέντε βουλευτέ οι οποίοι θέλουν να κάνουν ερωτήσει. Οπότε προτείνω να περιοριστείτε σε ένα λεπτό ο καθένα. Αλλιώ δεν θα ακούσουμε απαντήσεις. Ε, ε, uh, σας ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να σας ασκήσω λίγη κριτική γιατί ήταν πολύ ευγενικό, αλλά μετά στις απαντήσεις ε, ε, αποκαλύψατε τα διάφορα λάθη που έχει κάνει η Ευρώπη. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επεκταθείτε σε αυτό τον κατάλογο και να μας πείτε και τα υπόλοιπα λάθη που έχουν γίνει. Αλλά η πραγματική ερώτηση είναι πώς κρίνεται την προσέγγιση της Τρόικας στο ελληνικό πρόγραμμα, στο σχεδιασμό της ελληνικής ε, διεξόδου από την ε, κρίση, αν μπορείτε να μας ε, το περιγράψετε, γιατί είπατε πως εργάζονταν απομονωμένα, απομονωμένοι διάφοροι οργανισμοί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σάπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφερθήκατε στην οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίω. Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ινδία και στην Κίνα ε, ίσως να μην ε, έχουν τόσο μεγάλη σημασία γιατί βεβαίως βρίσκονται σε τελείως διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης από εμάς. Αλλά είπα βεβαίως είναι κάτι το διαφορετικό και είπατε πως ε, θα αυξηθεί τα επόμενα έτη το ΑΕΠ ε, της, τον είπα κατά 1% παραπάνω από ότι αυτό της Ευρώπης. Τι κάνει λοιπόν, τι κάνει οι Αμερικανοί καλύτερα από μας. Είναι κάτι το οποίο αφορά δημοκρατικούς παραγοντες, δημογραφικούς παραγόντες και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για τα δύο διαφορετικά δόγματα τα οποία συζητάμε συνεχώς είτε κάποια λιτότητα ή αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ οικονομία και δαπάνες από την άλλη. Αν δείτε το πώς εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε η κρίση, ποια είναι θα λέγατε η εμπειρία που μπορούμε να αντλήσουμε, πόσο βοηθάνε τα πακέτα ανάπτυξης δεδομένου του ότι εγώ θεωρώ πως ε, είχαμε ήδη πάρα πολλά κίνητρα γιατί ακριβώς ε, το έλλειμμα οφείλεται στις δαπάνες αυτές οι οποίες κατά την απόψή μου δεν απέδωσαν και το λέω και ήπια Σέρκο. Ευχαριστώ. Σύντομα θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, γνωρίζοντας το ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε ε, επενδύσει στην πραγματική οικονομία, ειδικά στην καινοτομία και στην ε, πράσινη ανάπτυξη. Και είναι ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι προτάσεις σας λοιπόν για αυτό. Σας ευχαριστώ. Άννη. Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί συνάδελφοι, κύριε Γενική Γραμματεία, έθεσαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και στις αρχικές σας παρατηρήσεις τονίσατε το ότι προσοχή πρέπει να δώσουμε στην πρόθεση της ανάπτυξης και της θέσης εργασίας και θίξατε το ζήτημα της εμπιστοσύνης, της εμπιστοσύνης των αγορών παρά το ότι εξίσου σημαντική είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών το ερώτημά μου είναι τι ακριβώς θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Ο σας ρώτησε για ε, τις ε, κύκλικες πολιτικές ε, σε χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα οικονομικής προσαρμογής όπως η Ελλάδα. Έχουμε τρία, και τα τρία αρνητικά και αυξάνονται οι ανισότητες και επιδεινώνεται η ύφεση και αυξάνεται η ανεργία. Καλές οι μεταρρυθμίσεις, αλλά χρειάζεται χρόνος για να δώσουν αποτελέσματα. Τι μπορούμε, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των πολιτών για να δημιουργηθούν οι όροι της επιτυχίας. Έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κρίση μου για την προσέγγιση της Τρόικας. Σαφώς η προσέγγιση αρχικά ήταν ότι ναι έχουμε εδώ πέρα ένα τυποποιημένο πρόβλημα ελλημάτων, το, τα ελλείμματα ήταν τεράστια. Εγώ θα το λέω λάθος εγκυλοποίησης γιατί μιλούσαν για 5% ενώ ήταν 15% αλλά καταλαβαίνετε πως το να μειωθεί αυτό το μέγεθος θα χρειάζεται βεβαίω πάρα πολλά χρόνια και χρειάζεται και ένα τεράστιο μέγεθος ΑΕΠ. Και ήταν και τιμωρητικά τα επιτόκια και το PSI ήταν ε, εντελώς μη ρεαλιστικό η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Χάσαμε λοιπόν δύο χρόνια με την Ελλάδα. Πριν δύο χρόνια έπρεπε να πούμε πως δεν τραβάει αυτή η κατάσταση. Όταν ήταν 300 δισεκατομμύρια το ιδιωτικό χρέος, όχι 200, 300 έπρεπε να πούμε 50% ή τέλος πάντων όσο θέλαμε. Τώρα επιτέλους ε, μειώθηκε μετά από 1,5 ε, χρόνο που πληρώναμε μετρητά 100 cents το ευρώ για, από τους φορολογούμενους σας στους ε, πιστωτές του ιδιωτικού τομέα. Και τότε συνειδητοποίησαμε πως δεν τραβάει άλλο η κατάσταση. Ε, αυτό ήταν το προπατορικό μας αμάρτημα. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για την αναδιάρθρωση. Δεν μπορούσαμε να προφέρουμε τη λέξη στο να απαγορευόταν. Γιατί το λέγανε και σας το μεταφέρω επί λέξη ανεύθυνο. Και ανεύθυνο και ανεύθυνο μας το είπαν. Τρεις φορές μου το είπανε, σαν τον Άγιο Πέτρο, πως δεν έπρεπε να ε, προφέρουμε αυτή τη λέξη. Στο τέλος, ε, ξεχάσανε πως ε, εγώ είμαι Μεξικάνος και είχαμε κάνει αναδιάρθρωση στη χώρα μου και δεν συνέβη τίποτα. Δεν ξανακοιτάξαμε ε, ποτέ πίσω, αναπτυσσόμαστε συνεχώς. Γιατί, γιατί χρησιμοποιείται το ευρώ και δεν μπορεί κανεί με το ευρώ να υπερδανιστεί, να κάνει λάθος, να χρεοκοπήσει, όχι. Δεν υπήρχαν αυτοί οι έλεγχοι όμω που θεωρούσατε ότι υπήρχαν και το επιτρέψατε να συμβεί. Ναι, αυτό θα γινόταν και με τη δραχμή και με το ευρώ και με το Μάρκο και με οτιδήποτε. Αν δανείζεται κανείς υπερβολικά δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του, 160% του ΑΕΠ έπρεπε να το έχετε αναγνωρίσει αυτό εξ αρχής. Αλλά χάσαμε το τρένο γιατί επί ένα έτος πληρώναμε πλήρως τους πιστωτές και λέγαν πως είναι ανεύθυνο να διανοηθούμε να πληρώσουμε κτλ. Τώρα η Τρόικα άλλαξε τελείως προσέγγιση, τους συγχαίρουμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά Χάσαμε την ευκαιρία. Να σας πω το εξής κυρία μου. Το κόστος του να λέμε δεν μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε, δεν μπορούμε να χρεοκοπήσουμε γιατί χρησιμοποιείται το ευρώ, η αβεβαιότητα όσον αφορά χρηματαγορές, αγορές αγαθών, απασχόληση, ανάπτυξη ήταν 50 έως 70 φορές το σύνολο του χρέους της Ελλάδας. Αυτό ήταν το κόστος. η Ευρώπη θα έπρεπε να πει αγοράζουμε όλο το χρέο τη Ελλάδα και θα το μοιραστούμε μεταξύ μα. Και θα ήταν 10 φορέ φτηνότερο από αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα. Γιατί, γιατί όχι δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε. Ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Πολύ κακή κατάσταση. Αλλά συνέβη τώρα, ελπίζω να μάθαμε και να είμαστε ρεαλιστέ. Ελπίζω να μην χρειάζεται να ξαναδούμε κάτι τέτοιο ποτέ, αλλά εάν χρειαστεί θα πρέπει να μάθουμε από αυτά τα λάθη. Τώρα για την Ινδία και την Κίνα και την ανάπτυξή τους ε, που λέτε πως δεν είναι τόσο σημαντική γιατί είναι σε διαφορετική φάση ανάπτυξης. Ναι, ε, το πρόβλημα είναι πως είναι τώρα οι μόνες χώρες που αναπτύσσονται. Η ΕΠΑ είναι για επισκευή και ο ευρωπαϊκός κινητήρας ανάπτυξης επίσης και η Ιαπωνία και ο μόνος κινητήρας που τραβάει όλη την οικονομία είναι αυτή. Και έχει διαφορά βεβαίω η ανάπτυξη του 11% από το 8% και το 7%. Εγώ θεωρώ καλύτερο να τίστε εκείνα στο 9% παρά στο 11% γιατί είναι πιο βιώσιμο. Απ' την άλλη, αν θα έχει αντίκτυπο στην ε, γενικότερη ανάπτυξη, ναι βεβαίω. Ε, ε, εννοείται, συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μαθηματικό είναι. Αλλά εάν και μια χώρα η οποία εξάγει, πού θα εξάγει, ποιο θα τα αγοράσει αυτά τα πράγματα. Εσεί δεν τα αγοράζετε, οι Αμερικάνοι δεν αγοράζουν, η Ιαπωνία δεν αγοράζει, Πώς περιμένετε η Κίνα και η Ινδία να αναπτυχθούν από μόνες τους, από την εσωτερική τους ζήτηση. Ναι, βελτιώνονται και εκεί, πρέπει να το πω, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Το ότι το εμπόριο έχει παγώσει ουσιαστικά, όχι έχει σταματήσει να αναπτύσσεται, είναι πολύ, σοβαρή, πολύ σοβαρό σύμπτωμα, αλλά ταυτόχρονα και αιτία του προβλήματος, γιατί ε, μετά επηρεάζει όλες τις μεγάλες χώρες ε, που εξάγουν. Τώρα, κύριε Χόκμαρκ, για τα δόγματα. Λιτότητα ή ανάπτυξη ή κίνητρα. Τα κίνητρα ήταν ε, κάτι το οποίο έγινε σωστά την στιγμή εκείνη, γιατί είχαμε μια τεράστια οικονομική κρίση. Μετά είχαμε οικονομική παράλυση σε όλο τον κόσμο, όταν ε, μεταδόθηκε σαν έμπολα η χρηματοοικονομική κρίση και μετά τι συνέβη. χρησιμοποίησαμε ό,τι περιθώριο υπήρχε στου προπολογισμού για να ξοδέψουμε, για να βγούμε από την κρίση. Αυτή ήταν καλή απόφαση. Εγώ την στηρίζω. Αυτό θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Όμω. αυτό έγινε από χώρε οι οποίε είχαν ήδη έλλειμμα 6% και χώρε όπω η Ισπανία που είχε πλεόνασμα. Ή χώρες ε, όπως η Γερμανία που είχαν μια ισορροπία. Η Γερμανία είχε περιθώριο, η Ισπανία είχε περιθώριο, ο Καναδά είχε περιθώριο και οι χώρες οι οποίες είχαν έλλειμμα 6% είχαν ελάχιστο περιθώριο και εξόδευαν 3-4-5% παραπάνω και ξέφυγαν εντελώς. Οπότε έχει περάσει τώρα η στιγμή των κινήτρων της κινητοποίησης της οικονομίας. Τώρα, το, οι επιλογές είναι, κοιτάξτε δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Ε, γιατί είναι και πολύ απλοϊκή αυτή η προσέγγιση. Το θέμα είναι το κατάλληλο μείγμα μεταξύ οικονομικής εξυγίανσης και τα στοιχεία εκείνα ανάπτυξη μπορούν να μπουν ακόμα και σε σφιχτό προπολογισμό. Εκπαίδευση, καινοτομία, πράσινη ανάπτυξη. Αυτά τα πράγματα θα μας ε, βοηθήσουν. Ξέρετε τι λέμε κύριε Χοκμάλ; Επειδή δεν έχουμε περιθώριο στην πολιτική, την νομισματική και του προπολογισμού, τα, τα επιτόκια είναι μηδέν, δεν πάνε παρακάτω, λέμε διαρθρωτικές αλλαγές κοινωνικά πράσινα. Αυτά λέμε. Αυτά λέμε στον ΩΣΑ. Διαρθρωτικέ αλλαγές. Τι εννοούμε. Εκπαίδευση, καινοτομία, ανταγωνισμός, έρευνα και ανάπτυξη, πανεπιστήμια, υγεία, φορολογία, κοινωνικά. Γιατί υπάρχουν 24 εκατομμύρια ανεργία αλλά και πολλά άλλα εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη που είναι θύματα της κρίσης και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό και πράσινη κατεύθυνση γιατί αν το δούμε και στην επόμενη γενιά είναι το, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε δεν νομίζω πως υπάρχει πως είναι ή το ένα ή το άλλο. Τώρα κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου και τι μπορούμε να κάνουμε για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Στην δημοσίευσή μας, ε, στοχεύοντας την ανάπτυξη που και πριν από λίγες εβδομάδες και σας καλώ να διαβάσετε, λέμε αυξημένος ανταγωνισμός ε, και δικτυωμένες βιομηχανίες. Ε, στήριξη στη Γεωργία, ζητώ συγγνώμη από όσους δεν τους αράσουν. Αυξημένος ανταγωνισμός στις υπηρεσίες, ε, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, αύξηση της κινητικότητας της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία αγορά, ενιαία αγορά, ενιαία αγορά. Αν τα κάνετε αυτά, Κοιτάξτε και εμείς τα ζητάμε αυτά από το 2007, 8, 9, 11 και του χρόνου. Πάλι μάλλον τα ίδια θα λέμε. Ελπίζω όχι, αλλά θα επιμένουμε. Και έτσι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, αύριο, επί τη ευκαιρία, αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά τυπώνονται, θα α, ε, μοιράσουμε εδώ πέρα στις Βρυξέλλες τις ε, οικονομικές μας έρευνες ε, και για την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Και σας ε, προσκαλούμε λοιπόν στην παρουσίαση της μελέτης αυτής για να δείτε τα τελευταία στοιχεία και τα νούμερα, αλλά η ουσία είναι αυτά τα οποία σας ανέφερα. Και για την εμπιστοσύνη σε χώρες με δημοσιονομικά προγράμματα προσαρμογής όχι, δεν θεωρώ πως ε, επειδή κάνετε δημοσιονομική προσαρμογή μπορείτε να ξεχάσετε τελείω την ανάπτυξη. Αλλά, αλλά, ας είμαστε ρεαλιστές. Κάποιες χώρες, τελείωσε ο χρόνος τους πριν από δύο χρόνια. Και κάποιες από αυτές τις χώρες το κατάλαβαν, κάποιες άλλες όχι. Και δεν ξεκίνησαν διαδικασία προσαρμογής πριν από δύο χρόνια. Έλεγαν, εμεί ε, είμαστε εμβολιασμένοι, δεν μα πιάνει η αρρώστια. Καθυστέρησαν άλλον ένα χρόνο για να ξεκινήσουν τη διαδικασία προσαρμογής. Και τώρα βλέπουμε ενάρετη συμπεριφορά, αλλά με δύο χρόνια καθυστέρηση, με ενάμιση χρόνο καθυστέρηση. Και το κόστος της προσαρμογής είναι πολύ υψηλότερο. Το τίμημα πλέον εισόδου είναι πολύ ακριβότερο. Η απόδοση των χωρών σήμερα για να ικανοποιήσουν την κρίση των αγορών που γίνεται όλο και πιο αυστηρή πρέπει να είναι πολύ πιο οδυνηρή, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι θα ήταν πριν από ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Με τη μισή προσπάθεια από αυτή η οποία απαιτείται σήμερα θα είχατε ικανοποιήσει τι αγορέ πριν από δύο χρόνια. Αλλά επειδή δεν έγινε, δεν πήραμε στα σοβαρά τι αγορέ, λέγαμε δεν μα καταλαβαίνουν οι αγορέ. Το πρόβλημα δεν, είναι, δεν υπάρχει κάποιο κύριο αγορά, κυρία αγορά. Οι αγορέ σα χτυπάνε όταν δεν σα πιστεύουν. Και ο μόνος τρόπος για να έχει κανείς αξιοπιστία είναι να ξεπεράσει αυτό το οποίο φαίνεται. Αν περιμένουν 50, δώστε τους 70, 100. Γιατί, γιατί έτσι μετά μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις. Αλλιώς, παραδείγματος χάρη, γιατί υπάρχει τόσο διαφορετικό αποτέλεσμα. Να δούμε την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα, και θα τελειώσω, μου λένε εδώ πέρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί ήταν αξιόπιστο. Ναι, και εντάξει, τώρα έχει λιγότερη ανάπτυξη. Γιατί παρουσίασαν ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξ αρχή και το τήρησαν. Γιατί κάποιες άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα δεν είναι τόσο αξιόπιστες. Γιατί έκαναν βηματάκι βηματάκι όπως τους ανάγκαζαν οι περιστάσεις. Δεν πέρασαν ένα τεστ αξιοπιστίας, αν θέλετε. Ήταν η στρατηγική Δεν ξεπέρασαν αυτό το οποίο χρειαζόταν. Λένε, εάν χρειάζομαι 100 και σήμερα σας δώσω 17, θα είναι ικανοποιημένες οι αγορές. Όχι. 23, μα σας δώσω όχι. Και κάθε φορά τα επιτόκια ανέβαιναν, ανέβαιναν. Και ειλικρινά, βλέπετε, τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να αναφέρω τα τετριμένα, η Γερμανία λοιπά, Ανέφερα δύο άλλες χώρες, Οι οποίε και οι δύο σήμερα δέχονται πίεση. Η μία ε, στον προπολογισμό, αλλά με πολύ καλή υποδοχή από τις αγορές και κάποια άλλη, οι οποία κάνουν πράγματα αλλά δεν τους πιστεύουν οι αγορές και δεν τους πιστεύουν γιατί επέλεξαν να το κάνουν σιγά σιγά και είναι πολύ οδυνηρό όταν σου κόβουν κομματάκι κομματάκι την ουρά. Μπορεί να την κόψουν μια, μια και καλή και να τελειώνει. Είναι ένα στρατηγικό ζήτημα. Και με αυτά τα εύθυμα, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, ε, πάντα χαίρομαι όταν κάθομαι δίπλα σας στο ΕΚΟΦΗΝ. Αλλά δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετιστούμε τώρα και θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξή μας. δηλαδή την, ε, ε, τις εκθέσεις του, των Ζωάν Πολ Γκοζές και Ελίζα Φερέιρα. Thank you. Jean Paul, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, σήμερα θα μιλήσω ιστανικά. Τι δεν προβλέπετε μετάφραση διερμηνία από εστονικά. Τρομερό. Τέλος πάντων, είχα αποφασίσει για ποικιλία να μιλήσω ιστονικά, λέει ο κύριος Γκοζές, αλλά θα μιλήσω γαλλικά παρόλα αυτά. Και συνεχίζεται η προσπάθεια και η μάχη. Έχουμε λοιπόν εγγεγραμμένα στη μέση διάταξη τη δικιά μου έκθεση και την έκθεση της ε, Ελίζα Φερέιρα. Θα μιλήσουμε πρώτα, αν μου επιτρέπετε και για λόγους ευκολίας, ε, για τη δικιά μου έκθεση, μετά για την έκθεση της Ελίζα, μετά σκιώδη κτλ. Θα μπορέσουν ε, οι ενδιαφερόμενοι να μιλήσουν για τη μία ή την άλλη έκθεση. Στόχος ε, λοιπόν ε, ε, του κανονισμού για να αντιμετωπιστούν δυσκολίες χωρών, οι οποίες είτε χώρες που είτε αντιμετωπίζουν οι δυσκολίες είτε φαίνεται ότι θα τις αντιμετωπίσουν όσον ο νούπο, αφορά την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής τους εποπτείας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο ζήτημα αυτό έχει ήδη πάρει ε, το ΕΚΟΦΗΝ εδώ και πάνω από ένα μήνα και η συζήτηση λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ε, δεν είναι βέβαια απλό ζήτημα. Οι συνάδελφοι δε έχουν ήδη ε, υποβάλει σειρά τροπολογιών, 200 τροπολογίες περίπου για το δικό μου κείμενο ποια είναι τώρα τα σημεία τα οποία ε, προκαλούν περισσότερα προβλήματα ή ποια είναι τα σημεία τα οποία αξίζουν περισσότερη συζήτηση. Εξ αρχής διαπίστωσα στο κείμενο της ε, Κομισιόν ότι αποφάσιζε μόνη τη, ε, χωρί να γίνεται ποτέ λόγος ή σχεδόν ποτέ λόγος για το Συμβούλιο όσον αφορά την απόφαση εποπτεία για τα πρώτα μέτρα. Έξεπλάγει από την κατάσταση αυτή έμαθα δε ότι είχε γίνει μεγάλη συζήτηση στο Συμβούλιο ε, και ότι αποφασίστηκε ότι τελικά οποιαδήποτε αναφορά στη θέση της, ε, του Συμβουλίου ε, δεν θα ανεφέρω Κατά την άποψή μου δεν είναι πολύ συνεκτικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όποιος και είναι ο βαθμός παρέμβασής της, να μπορεί λέω να παίρνει αποφάσεις χωρίς οποιαδήποτε στιγμή το Συμβούλιο να παρεμβαίνει. Βεβαίω μπορούμε να πούμε ότι αυτό δίνει ανεξαρτησία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνει της δίνει και τη δυνατότητα να ενεργήσει, αλλά νομίζω νομίζω ότι αυτή τελικά η ελευθερία ενέργειας μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι ε, γιατί μπορούν να πιέσουν τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε αυτή να μην πάρει μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω εξ αρχής ε, να μπορούν να απορριφθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Συμβούλιο, από εντεστραμμένη πλειοψηφία. Θα δούμε αν θα είναι απλή ή ενισχυμένη η συζήτηση με τους συναδέλφους, ενδεχομένως θα μας επιτρέψει να πάρουμε μια πιο θέση. Η απλή πλειοψηφία θεωρήθηκε ότι ε, ίσως ε, δεν θα πρέπει να επιλεγεί και κατά αναλογία με το six pack να επιλέξουμε την ε, ενισχυμένη πλειοψηφία. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η ταύτιση με την περίφημη αυτή διακυβερνητική συμφωνία ή συνθήκη και εκφράστηκε η άποψη ότι ενδεχομένω θα μπορούσε να ενταχθεί στο κείμενό μου, ε, να ενταχθούν μάλλον κάποιες διατάξεις αυτής της διακυβερνητικής ε, συμφωνίας που θα μπορούσαν να εγγραφούν στο δεύτερογενέ δίκαιο, χωρίς βεβαίως να μπούμε ε, στην ουσιώδη ιδιαιτερότητα της διακυβερνητικής συνθήκης, δηλαδή του χρυσού κανόνα, έτσι όπως αποφασίστηκε από τα κράτη-μέλη. Αυτό το ζήτημα θα το αφήσουμε στην συνθήκη που εγώ ξέρετε ότι ονομάζω συμφωνία μετόχων. Ε, υπάρχει και ένας νεοτερισμός, ε, δηλαδή αυτός ο καθορισμός ενός ε, συστήματος πολύ δύσκολης εποπτείας, βλέπε προστασίας ενός κράτους που αντιμετωπίζει δυσκολία. Πιστεύω ότι αυτή είναι η λογική συνέπεια και συνέχεια των διαφόρων μέτρων που θα έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εις περίπτωση κατά την οποία δεν θα έχουν τα μέτρα αυτά οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτοί που είναι κατά του σχεδίου αυτού ε, λένε ότι με τον τρόπο αυτό θα ε, μπορούσαν τα κράτη να, ε, βάλουν, να δημιουργήσουν ένα σύστημα το οποίο θα τους, θα τους ξέπλαινε από κάθε ευθύνη τη στιγμή που θα έμπαιναν πλέον σε ένα καθεστώς εποπτείας. από την άλλη πλευρά βεβαίως προστατεύεται το κράτος σε περίπτωση κατά την οποία επαναλαμβάνω και τονίζω τα μέχρι τότε προτινόμενα μέτρα δεν θα έχουν δώσει αποτέλεσμα και εάν και εφόσον τα, τα, κράτη αυτά θα βρίσκονται ένα βήμα πριν την πτώχευση, τη στάση πληρωμών. Ε, έχω λάβει υπόψη μου πάρα πολλά στοιχεία και αντιρρήσεις ε, γιατί ε, υπάρχει έτσι μια μεγάλη σειρά αντιρρήσεων που ε, έχουν ακουστεί. Αυτό το σύστημα της ενίσχυσης της οικονομικής δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών θα μπορούσε να καλύψει, να προστατέψει τις χώρες από την άμεση ε, απειλή, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα τα οποία θα έχουν προταθεί ε, και θα έχουν συμφωνηθεί από την Κομισιόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφενός και την ενδιαφερόμενη χώρα από την ε, υπάρχει το Chapter 11 στις ΗΠΑ από το οποίο θα μπορούσαμε ε, να εμπνευστούμε. Δηλαδή πρώτα απ' όλα ενδεχομένως ε, ένα πάγωμα πρώτης, πρώτου παγώματος της, του χρέους, μετά ένα credit event, ένα πιστοτικό γεγονός το οποίο θα είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση απέτηση πληρωμής και μετά το ξεπάγωμα ας πούμε των χρεών της χώρας αυτής. Ε, μία άλλη οδός θα μπορούσε να ήταν ε, η εξυγίανση των οικονομικών ε, μετά από μία χρονική, χρονικό περιθώριο το οποίο θα έχει συμφωνηθεί. Η πρώτη πρόταση είναι ότι στην ουσία με τον τρόπο αυτό δεν, δεν δίνεται αξιοπιστία στους πολιτικούς που λένε ότι αυτό που είδαμε στην Ελλάδα δεν πρέπει να το ξαναδούμε. Άκουσα μόλις ε, τον πρόεδρο του ΩΣΑ ο οποίος ε, ενδιαφέροντα πράγματα μας είπε ε, και βεβαίως και μας είπε ότι δεν θα πρέπει να πάρουμε έτσι σαν δεδομένα τα, τα στοιχεία. Γιατί από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κατά τη δεν, δεν διώχνουμε την αρρώστια όταν οικοδομούμε ένα νοσοκομείο, αλλά τη στιγμή που αρρωσταίνουμε το νοσοκομείο καλό είναι να είναι κοντά μας. Δεύτερον, από τη στιγμή που υπάρχει ένα σύστημα προστασίας, αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποια στιγμή ε, θα μπορούσε να πτωχεύσει μια χώρα, να κάνει στάση πληρωμών και να μην μπορέσει να πληρώσει τις ε, υποχρεώσεις της. Ε, και επομένως η χώρα αυτή μέσω αυτών των συστημάτων έχει τη δυνατότητα να ανακάψει. Και αυτό που είπε προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, εάν τον κατάλαβα καλά, είναι ότι αν είχαν ληφθεί κάποιες αποφάσεις 1,5 2 χρόνια πριν, ε, ακόμα και αυτό της ε, πλήρους αναδιάρθρωσης ε, ή εξαγορά τέλο πάντων του ελληνικού χρέους δεν θα χρειαζόταν τώρα να πάρουμε τόσο σοβαρά μέτρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μου λένε καμιά φορά επικρίνοντας την εργασία μου ότι ξέρετε κάτι θα δημιουργήσετε μεγάλη ε, ε, μεγάλο φόβο στις αγορές. Μα όχι, καθόλου. Βεβαίως η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε σταθερή ε, πορεία και να προβλέπουμε τις καταστάσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι οι αγορές είναι ικανοποιημένες όπου για 1,5-2 χρόνια δεν ξέρουν ε, δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπιστούν ας πούμε οι πιστωτές της Α ή της Β ή της Γ χώρας, είναι καλύτερο αυτό. Ε, νομίζω ότι αυτά τα επιχειρήματα δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά γιατί από τη μία πλευρά δεν μπορούμε ε, να πούμε με τα απολύτους ευεβαιότητος ότι ποτέ ξανά καμία χώρα δεν θα αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία, στην Ισπανία και άλλες χώρες και από την άλλη πλευρά Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί ένα ε, σαφές νομικό καθεστώς το οποίο να διευκολύνει τις λύσεις και από αυτού θα συμφωνήσουμε όλοι, επί του συστήματος δηλαδή. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίω να υπάρχει σαφή διασύνδεση ανάμεσα σε αυτό το προτινόμενο νομικό σύστημα υποπτία κτλ. και ε, τη δημοκρατική λειτουργία του κράτου αφετέρου. Θα πρέπει να βρεθεί και ομολογώ ότι ακόμα δεν έχω καταλήξει, περιμένω και τι σκέψει που θα εκφράσουν οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα το οποίο να είναι αποδεκτό, το οποίο θα επιτρέπει ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των προτινόμενων μέτρων που θα ε, διαπραγματευτεί η χώρα, η νόμιμη εκπρόσωπος δηλαδή, ε, της, ε, ε, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της χώρας που θα συμφωνήσουν για την ανόρθωση της χώρας με τους πιστωτές και θα πρέπει μέσα σε πλαίσια δημοκρατικού διαλόγου και δημοκρατικών διαδικασιών να γίνονται όλα αυτά. Αυτά είναι τα προβλήματα που με απασχολούν σήμερα. Ευχαριστώ βεβαίως όλους τους συναδέλφους που έχουν ήδη προτείνει κάποιες τροπολογίες. Έχω ήδη συνεργαστεί με τους σκιώδεις εισηγητές ε, και έχω ήδη καταλήξει σε κάποια προσχέδια διατύπωσης. Ε, ακόμα έχουμε βέβαια πολλή δουλειά μπροστά μας. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να γρηγορούμε. Και επιμένω και ότι το ΕΚΟΦΗΝ ήδη έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Εάν θέλουμε το Κοινοβούλιο να ε, συμβάλλει με μία σειρά συγκεκριμένων αυτών ε, ιδεών, ε, θα πρέπει να γρηγορήσουμε, θα πρέπει γρήγορα να, να μιλήσουμε, θα πρέπει γρήγορα να ακουστεί η φωνή μας, γιατί διαφορετικά θα αποδυναμωθεί αυτή η φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε η Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον ε, κύριο Κοζές για το έργο που έφερε σε πέρας ως εισηγητής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να εξασφαλίσει τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές μέσα σε ένα πνεύμα διαλόγου και με συμπερίληψη όλων των απόψεων. Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Κοζές, Πιστεύω ότι αυτό το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή. Γιατί? Γιατί είναι πια σαφές ότι δεν είναι μονάχα η εφαρμογή του η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια ταξινόμηση των χωρών. Μπορεί πραγματικά να καταταγεί μια χώρα σαν μια χώρα που είναι πολύ κοντά στην αφαιρεγγιότητα αλλά επίσης και γιατί δίνει τη δυνατότητα στις υπόλοιπες χώρες οι οποίες βρίσκονται μέσα στη ζώνη του ευρώ να υποχρεώσουν μια χώρα να προσφύγει στη βοήθεια των υπολείπων, ουσιαστικά λοιπόν να προκαλέσουν μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτή που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Είναι ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο είναι από τη φύση του ήδη πάρα πολύ πολύπλοκο και του οποίου οι συνέπειες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή και επιφύλαξη. Εγώ έχω προτείνει μια σειρά από τροπολογίες οι οποίες έχουν σαν στόχο να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ όλης αυτής της διαδικασίας και των απορριών της και της προηγούμενης κατάστασης η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί όταν εμείς ξεκινάμε μια νομοθετική διαδικασία η οποία έχει τόσο σοβαρές συνέπειες. Αυτό λοιπόν που προτείνω με τις τροπολογίες μου και ιδίως με την τροπολογία 104 είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια βαθμία διαδικασία ώστε να μπει μια χώρα στη διαδικασία αυτή της ενισχυμένης εποπτείας όταν η χώρα αυτή ήδη βρίσκεται στη διαδικασία επισκόπησης του χρέους της λόγω μακροοικονομικών ανισοτήτων και όταν συνεχίζει αυτή η διαδικασία και μπαίνει στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Επομένως, εγώ θα ήθελα να υπάρξουν συνδέσεις μεταξύ του μηχανισμού ο οποίος έχει ήδη ε, προετοιμαστεί στα πλαίσια του ΣΥΚΠΑΚ της εξάπτυχου, ώστε να μην θεωρείται ότι μια χώρα μπορεί να μπει σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι προθάλαμος της αφαιρεγγιότητος χωρίς να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι έχουν θεσπιστεί στο παρελθόν ώστε να κατευθύνουν τη διαδικασία παρακολούθησης μιας χώρας που εμπλέκεται στην λεγόμενη ενισχυμένη υποπτία. Γι' αυτό η τροπολογία μου, η 104, προτείνει να υπάρχει μια δυτή προσέγγιση, μια μορφή προσέγγισης όπου ζητείται από μια χώρα ένα σύνολο πληροφοριών, αλλά η οποία ανταποκρίνεται σε ένα πιο ελαφρό επίπεδο παρακολούθησης, δηλαδή όταν μια χώρα προσυπόκειται σε ενισχυμένη παρακολούθηση, που είναι αποτέλεσμα του ελέγχου του κρατικού χρέους, και μια δεύτερη διαδικασία όταν μια χώρα έχει ήδη ζητήσει την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου Πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί σε σχέση με τις πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να ζητούνται από τη χώρα αυτή. Αυτές είναι λοιπόν η τροπολογία 128, 130, 133, 134 και 420. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η σχέση μεταξύ αυτού που προτείνεται εδώ και αυτού που έχουμε επιτύχει στην, στο, στο εξάπτυχο νομοθέτημα, στο six pack, είναι σε σχέση με τις συστάσεις που υποβάλλονται προς μια χώρα να μην είναι ασυνάρτητες αυτές, να μην υπάρχουν κάθε μορφή συστάσεις, να υπάρχει μια συνεκτικότητα. Αυτό το οποίο ζητείτε λοιπόν από μια χώρα ότι πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός προγράμματος όταν βρίσκεται κάτω από πιο στενή εποπτεία, όταν βρίσκεται υπό ενισχυμένη εποπτεία, όλα αυτά λοιπόν τα οποία ζητούνται από τη χώρα αυτή θα πρέπει να είναι συμβατά και να συνάπτονται με αυτά τα οποία προβλέπονται από το Σύμφωνο Σταθερότητος και από τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταρρύθμισης. Δεν είναι λοιπόν επειδή μια χώρα βρίσκεται σε πιο δύσκολη κατάσταση ή σε πιο ε, επισφαλή θέση ότι μπορούμε να ξεχάσουμε όλες τις προηγούμενες συστάσεις και να κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχει επίση και ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω από πολιτική έποψη, είναι το πρόβλημα το οποίο προκύπτει όταν μια χώρα η οποία έχει φτάσει σε μια κατάσταση που είναι υποχρεωμένη να ζητήσει βοήθεια, ουσιαστικά αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πιέζεται από τις άλλες χώρες της ζώνη του ευρώ, αλλά δεν έχει την δυνατότητα να δώσει μια θετική απάντηση σε αυτό το αίτημα, διότι δεν καλύπτεται από το σύστημα σταθερότητας ή τα μελλοντικά συστήματα σταθερότητας. Και το λέω αυτό στην τροπολογία 144, ότι εάν μια χώρα υποχρεώνεται να προχωρήσει στην αίτηση αρρωγής, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται αυτό από μια εγγύηση ότι θα τύχει πράγματι αυτής της αρρωγής, γιατί αλλιώς την αφήνουμε στο έλεος των αγορών. Ε, για αυτά που είπε ο κύριος Γκοζές επίσης. Δεν θέλησε ο κύριος Γκοζές να εισαγάγει μια ορολογία η οποία προέρχεται από την ε, διακυβερνητική συμφωνία το σύμφωνο αυτό, αυτό ήδη ένας καλός ε, ιονός. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει να έχουμε ένα ισορροπημένο κείμενο στο τέλος. Και υπογραμμίζω επίσης θετικά ότι ο κύριος Γκοζές αναφέρθηκε σε αυτή την έννοια του κεφαλαίου 11, σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα των ΗΠΑ. Να υπάρχει λοιπόν μια τέτοια διαδικασία, νομίζω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα που αξίζει να την διερευνήσουμε και να μπορέσουμε, ελπίζω ότι με καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλικομένων μπορούμε να φτάσουμε σε μια πιο ισορροπημένη λύση, γιατί νομίζω ότι αυτή ήταν πράγματι η ιδέα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος. Έχουμε περίπου μια ώρα στη διάθεσή μας και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ο Καρλ έχει να λάβει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Sharon. Κάποιες σκέψεις από πλευράς φιλελευθέρων. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί ήταν πάρα πολύ επικοδομητικός και είχαμε μια συζήτηση σε καλή ατμόσφαιρα. Νομίζω πως Βασικό στόχο η ομάδα μας εδώ πέρα έχει να ενισχύσει την επιτήρηση και τη δυνατότητα παρέμβασης ε, πριν ε, γίνουν απολυφιστικά τα προβλήματα και βεβαίως ε, προς τα εκεί στοχεύουν οι τροπολογίες μας. Τις περισσότερες έχω υποβάλει εγώ με τη στήριξη της ομάδας. Ένα από τα ζητήματα που καλύπτει ε, πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε αφορά τη συμπεριφορά στις ψηφοφορίες στο Συμβούλιο και το έχουμε πει πολλές φορές στο εξαπλό αυτό πακέτο καθώς είχαμε πολλά παζάρια στο Συμβούλιο και θεωρούμε πως θα πρέπει να επιλέξουμε μια λύση με αντιστραμμένη ειδική πλειοψηφία για να είμαστε σίγουροι πως θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις όταν χρειάζεται. Κατόπιν όταν ε, πρόκειται για την ε, πρώτη απόφαση μιας χώρας ε, σε ενισχυμένη εποπτεία θα πρέπει να ξέρουμε πως στο πλαίσιο αυτό ούτε και το Συμβούλιο είναι κατά της πρότασης της Κομισιόν. Υπάρχει αυτή η διαδικασία εντός του εξαπλού πακέτου, οπότε είναι φυστάμενη για το πώς θα πρέπει να εποπτεύει η Κομισιόν την κατάσταση πριν προχωρήσει σε μέτρα. Αυτό είναι φυσικό. Ποτέ δεν έχουμε ορίσει το τι σημαίνει αυτή η μελέτη μιας χώρας σε βάθος, αλλά είναι φυσικό η Κομισιόν να μην ε, θέτει κάποιον υπό ενισχυμένη υποπτία χωρίς να υπάρχει λόγος. Οπότε θα θέλαμε να αλλάξει το η πρόταση της Κομισιόν για το τμήμα αυτό της διαδικασίας. Επίσης, θέσαμε μια πρόταση και λέμε πως για να είναι πιο ισχυρή η εποπτεία θα είναι υποχρεωτική η λήψη αποφάσεων από την Κομισιόν αντί για τον αρχικό προαιρετικό χαρακτήρα που θα είχαν. Κατόπιν έχουμε καταθέσει και άλλες κάποιες προτάσεις στο άρθρο 6 3 για να αυξηθεί η δυνατότητα άσκησης πίεσης στα κράτη-μέλη που δεν ε, θέλουν να συνεργαστούν στο πρόγραμμα μακροοικονομικής ε, προσαρμογής κατόπιν όσον αφορά το ζήτημα του κεφαλαίου 11. Νομίζω πως οι περισσότεροι βουλευτές της ομάδας μας βλέπουν το σκεπτικό, αλλά το θέμα είναι αν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να εισαχθεί μια τέτοια λογική π.χ. Ο μόνος λόγος τον οποίο θα μπορούσα εγώ να δω είναι οι χώρες, ε, οι νότιες ε, της Ευρώπης ε, θα καταλήξουν να χρεοκοπήσουν επειδή δεν τους εμπιστεύονται οι αγορές. Δεν ξέρω λοιπόν πως, δεν ξέρω αν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να στείλουμε το μήνυμα πως υπάρχει και η πιθανότητα της χρεοκοπίας. Οπότε έχουμε κάποιες επιφυλάξεις απέναντι σε αυτό. Αν και δεν λαμβανόμαστε πως μακροπρόθεσμα είναι απαραίτητο, απλά ε, δεν ξέρουμε αν τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για το λεπτό αυτό θέμα. Κατόπιν, για το ζήτημα ενσωμάτωσης του Δημοσιονομικού Συμφώνου στους δύο κανονισμούς, έχουμε καταθέσει τροπολογίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή της ε, ε, πολιτικής ένωσης ε, για τα διαρθρωτικά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να στείλουμε το μήνυμα ότι επιτρέπουμε ένα ε, έλλειμμα 0,5% αντιλαμβάνομαι βεβαίως τα του συμφώνου αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε πράγματι τέλος μια που λείπει ο συντονιστής μας ή η συντονιστρια μας να πω κάποια πράγματα εξ ονοματός της. Πρώτα απ' όλα η Σίλια λέει πως θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ του εξαπλού πακέτου και εγώ συμφωνώ μαζί της για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα παραθυράκια αλλά και για να λειτουργεί η διαδικασία από πλευράς κομισιών όταν θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα που δημιουργούμε. Κατόπιν η Σίλια Θέλει να πει πως δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέοι ριζοσπαστικοί μηχανισμοί που μπορούν να δημιουργήσουν και παρεξηγήσεις. Και στην κατάσταση στις ε, χρηματαγορές και νομίζω πως αναφέρεται σε αυτό που είπα και εγώ πριν για το κεφάλαιο 11 μετά, η ομάδα μας θέλει να τονίσει πως το Ταμείο Διάσωσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να θίξουμε εδώ πέρα. Γιατί κατά την άποψή μας είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος αντιμετώπισης ε, της ε, κρίσης και θα το θα το βρούμε μπροστά μας παρά τα καλύτερα μηνύματα από τις αγορές ε, εσχάτως. Τέλος, η Σίλια θέλει να τονίσει πως τα κράτη-μέλη ε, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες... Ε, Α, όχι, τι διαβάζω. Όχι, όχι, αυτό αφορά τη φοροδιαφυγή, ναι. Θέλει να θίξει το ζήτημα της φοροδιαφυγής αν μπορούμε να το δούμε σε αυτό το πλαίσιο. Και ευχαρίστω να την στηρίξω. Αυτά από εμένα και εξ ονόματος της ε, συντονίστριας. Σας ευχαριστούμε και αν... Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να τονίσω πρώτα απ' όλα πως στηρίζω τις ε, πρωτοβουλίες ενισχυμένης οικονομικής ε, διακυβέρνησης Ευρωζώνης. Ε, με επικοδομητικό πνεύμα λοιπόν κατέθεσαν τροπολογίες και στην έκθεση Γκοζέ και στην έκθεση Φερέιρα και θα τονίσω κάποιε από αυτές σήμερα. Στην έκθεση Γκοζέ ήδη ανέφερα στην τελευταία μας συζήτηση στην Επιτροπή μας πως μπορούμε να στηρίξουμε πολλέ από τις προτάσεις του κυρίου Γκοζές. Χαίρομαι για το ότι αυτό συνεχίζει να ισχύει για πολλέ από τις συμβιβαστικές τροπολογίε. Στην τροπολογία μου υπαριθμών 180 τονίζω την σημασία του να αποφευχθεί η διπλή υποχρέωση υποβολής αναφοράς των κρατών μελών που βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Συμφωνώ με τον κύριο Γκοζές πως θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα νομικής ε, προστασίας ε, όπως ισχύει για τις περιπτώσεις χρεοκοπίας για τα κράτη αυτά. Η τροπολογία μου 229 λέει πως εάν ένα κράτος μέλος δεν θέλει να παραδώσει την δημοσιονομική του κυριαρχία πρέπει να έχει την επιλογή να βγει από την Ευρωζώνη. Η Κομισιόν και το Eurogroup θα πρέπει να βοηθήσουν τότε το εν λόγω κράτος μέλος με πρακτικά βήματα για να καταστήσουν την αποχώρηση από την Ευρωζώνη εφικτή και όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Στις ε, τροπολογίες μου, τώρα μιλάω για την έκθεση Φεραίρα ε, τις 65 και 192 στην έκθεση Φερέιρα, προτείνω σχέδια έκδοσης ομολόγων να αποτελούν επίσης μέρος του προϋπολογισμού που υποβάλλει το κράτος μέλος στην Κομισιόν για την διαδικασία αυτή και αν αναγκαίο η Κομισιόν θα ε, εκδώσει μια γνωμοδότηση για το σχέδιο προϋπολογισμού του κράτους μέλους με στόχο να αξιολογήσει το εάν οι συστάσεις που έγιναν προς το κράτος μέλος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αντιμετωπίστηκαν επαρκώς. Στις τροπολογίες μου 93 και 217 προτείνω πως η Κομισιόν θα πρέπει να αιτιολογεί όλες τις συστάσεις της για προσαρμογή του Εθνικού Προπολογισμού ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, το Εθνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση με απλή πλειοψηφία να αποφασίσει το εάν η γνωμοδότηση αυτή δεσμεύει τον λόγο κράτους μέλος ή όχι. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των προτινόμενων μέτρων. Σε απαιτήσει δημοσιότητας ε, τονίζω στροπολογίε 2.17 και 2.23 πως η γνωμοδότηση της Κομισιόν πρέπει να είναι δημόσια στο σύνολό της, εάν, εκτός εάν η Κομισιόν μετά από την σύμφωνη γνώμη του Eurogroup αποφασίσει αλλιώ το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις αξιολογήσεις της συνολικής δημοσιονομικής κατάστασης και προοπτικές της Ευρωζώνης στο σύνολό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντέρκ. Νομίζω ότι έχει σχολιάσει και την έκθεση της Ελίζα. Εντάξει, το επιτρέπω αυτό γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά να επανέλθουμε στην έκθεση του Ζωάν Πολ, δίνω το λόγο στο Σβέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία ελέγχθηκαν ήδη. Οι δικές μας τροπολογίες δείχνουν ότι καταρχήν υποστηρίζουμε τη βασική προσέγγιση της Κομισιόν να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια για τον τρόπο αντιμετώπισης των χωρών οι οποίες έχουν δυσκολίες σε σχέση με το οικονομική τους κατάσταση. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ασφάλεια σε νομικό επίπεδο και επίσης να φαίνεται και ο δημοκρατικός χαρακτήρας της λήψης αποφάσεων για αυτά τα μέτρα. Και αυτό ήταν και ο στόχος της, του κανονισμού αυτού. Επίσης υποστηρίζουμε να υπάρξει, να υπάρξει και μείωση του άχθους που προκύπτει από παράλληλες διαδικασίες όπως γίνεται τώρα. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν εκθέσεις προς την Τρόικα, διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος, διαδικασία λογανισόμεριων, όλες συμπούρμπουλες οι διαδικασίες αυτές μαζί με παράλληλους μηχανισμούς κυρώσεων. Όλες αυτές οι διαδικασίες λοιπόν θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους, αλλά διατηρώντας την ανάγκη να δίδονται εκθέσεις και να υπάρχει μια αξιολόγηση των ανισομεριών και ελλείψεων ισορροπιών που παρουσιάζουν. Επίσης οι τροπολογίες μας προτείνουν ότι θα πρέπει να επιτύχουμε και μια επανεξισορρόψη σε διάφορα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, όταν είναι δυνατόν, οι προτάσεις του Δημοσιονομικού Συμφώνου θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στο κείμενο αυτό και αυτό είναι και μια ευκαιρία πιστεύω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναφέρει στο ενωσιακό πλαίσιο διαδικασίες που είναι τώρα μονάχα διακυβερνητικές. Πάρα πολλά από αυτά λοιπόν βρίσκονται στην έκθεση της Ελίζα, αλλά πολλά άλλα στην έκθεση του Ζαν Πολ και νομίζω ότι είναι στο συμφέρον όλων των κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει ουσιαστικά επανενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο όλων αυτών των στοιχείων που έχουν να κάνουν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και την Διακρατική Συμφωνία. Αυτή είναι και η θέση που ανέφεραν οι φιλελεύθεροι. Επίσης, για το Ταμείο ε, απόσβεσης. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ήδη υπάρχον, το ιστορικό χρέος. Αυτά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε και είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα ταμείο απόσβασης και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει κάποιος τρόπος απορρόφησης και ακύρωσης του παλαιού χρέους. Σε σχέση επίσης με την αξιολόγηση των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής στις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, θα πρέπει να υπάρξει πλήρη συμπερίληψη και των κανόνων αξιολόγησης της Ευρώπης 2020. Θα πρέπει να έχουν λοιπόν σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, να ληφθούν υπόψη και τα αρνητικά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να προκληθούν από την εφαρμογή αυτών των κανόνων, ακόμα και τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να προκύπτουν από την εφαρμογή ενός προγράμματος σε μια άλλη χώρα. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε μια μονοκόμματη αντιμετώπιση ότι μια χώρα που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση μπορεί να προξενήσει αρνητικά προβλήματα σε άλλες χώρες και επίσης το γεγονός ότι όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή για ορισμένε από τις χώρες που έχουν προβλήματα ότι η κατάστασή τους μπορεί να οδηγήσει σε ένα κύμα φοροδιαφυγής και φυγής κεφαλαίων. Θα πρέπει η Ευρώπη να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και τέτοια προβλήματα. Μία ακόμα αρχή την οποία προσπαθούμε να εισαγάγουμε με τις τροπολογίες μας, είναι ότι απαιτείται πολύ περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των χωρών που βρίσκονται σε κρίση. Δεν είναι θετικό τελικά, δεν είναι προς όφελος των χωρών αυτών να δημοσιεύονται σημαντικά έγγραφα από τους Financial Times ή από άλλα έντυπα. Υπάρχει ένα είδος τρόμου που προξενείται από την διαρροή και δημοσίευση αυτών των εγγράφων. Και αυτά μπορεί να οδηγήσουν και σε κάποια αρνητικά αποτελέσματα στις ε, αγορές. Αν αυτά τα έγγραφα δημοσιεύονται με έναν τρόπο ο είναι συνεκτικός και διάφανος, θα είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα και πιστεύουμε ότι η κάθε χώρα έχει δικαίωμα πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα τα οποία την αφορούν και που περιλαμβάνουν τις αποστολές που αναφέρει ο κανονισμός ότι πρέπει να λάβουν χώρα και επίσης σε σχέση με την έννοια του βιώσιμου ή μη βιώσιμου χρέους για κάθε χώρα. Και αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να προετοιμάζονται λαμβάνοντας υπόψη και το, την θέση των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά είναι αξίες και αρχές που ακολουθούνται πλήρως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα για τέτοιες περιπτώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υπολείπεται των αρχών οι οποίες ισχύουν και πριτανεύουν στις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους εταίρους. Θα πρέπει να υπάρχει ο μέγιστος βαθμός διαφάνειας σε σχέση με αυτά τα οποία δημοσιεύονται. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο λοιπόν, αλλά θέλω να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια ευρεία συνένεση για τα ζητήματα αυτά και όλος ιδιαίτερος ο κανονισμός για τις χώρες που βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία θα πρέπει να τον δούμε με μια θετική αντιμετώπιση γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπιστήκανε στην ε, εξάπτυχο το ΣΥΚΣΠΑΚ, έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να δημοκρατικοποιήσει περισσότερο τις διαδικασίες αυτές και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι μας παρακολουθούν από πολύ κοντά για να δουν αν θα πάρουμε στα σοβαρά όλα αυτά τα προβλήματα. Κάποιες από τις προτάσεις λοιπόν του Ζωάν Πολ και από άλλους συναδέλφους είναι πολύ ελπιδοφόρες. Μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία γίνονται τώρα στις αποστολές της Τρόικα στις διάφορες χώρες. Ο Νικόλας Χούντης έχει το λόγο. έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εισηγητών μας, θα αναφερθώ κυρίως στην έκθεση του κυρίου Γκοζές, δεν μας έπεισαν ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση σε σχέση με τους δύο κανονισμούς. Η στάση μας είναι αρνητική. Συμπυκνώνεται στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί 47 και 48 και από εμά και από δύο σοσιαλιστές που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να απορρίψει τις προτάσεις της Επιτροπής. Και το οφείλει είναι ότι κάποια στιγμή αυτός ο παροξισμός αυτών των μέτρων πρέπει να πάρουν ένα τέλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη γνώμη μας πρέπει να πείτε ότι τις απορρίπτει αυτές τις προτάσεις. Όσο αφορά εμάς και στην προφορική συζήτηση αλλά και όταν συζητούσαμε και το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης που οι δύο νέοι κανονισμοί θέλουν να το κάνουν ακόμα πιο αυστηρό είχαμε εκφράσει τη ριθιστική μας διαφωνία και γιατί ήταν λάθος απάντηση στα κρισιακά φαινόμενα ή στην πρόληψη της κρίσης, αλλά γιατί και τώρα πολύ περισσότερο τα αποτελέσματα μιας τέτοιας πολιτικής ήδη είναι πολύ ορατά. Είναι τα αποτελέσματα στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία με τα στοιχεία που βλέπουμε, στην Ισπανία ενδεχομένως και που θα έχουμε την ευκαιρία αναλυτικά αύριο στην καταπρόσωπο ας το πούμε έτσι συζήτηση με την Κρόικα, Τρόικα να δούμε τι συνταγές είναι αυτές και τι αποτελέσματα βγάζουν. Επομένως έχοντας αυτή την εικόνα συμφωνούμε ότι και από οικονομική και από πολιτική άποψη αυτές οι προτάσεις πρέπει να απορριφθούν. Κατά τα άλλα για να μην ε, καταχρώμε του χρόνου ε, σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Κοζές, επειδή στην προηγούμενη πρώτη συζήτηση είχε αφαιθεί μια σύγχυση ε, από δική μου ή δεν είχε, ε, ας το πούμε έτσι, αποδοθεί σωστά, είμαι σύμφωνος. Είμαι με την τροπολογία 3, δηλαδή ότι πρέπει να διαγραφούν οι προβλέψεις, ότι πρέπει μια χώρα η οποία είναι απίθαρχη ανάμεσα στις άλλες κυρώσεις και τιμωρίες να περιορίζονται, να κόβονται οι ροές από τα ταμεία συνοχής. Από αυτή την άποψη με τον εισηγητή συμφωνώ και το, ας το, πούμε, το διευκρινίζω τώρα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ε, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, που πιο ε, συγγνώμη, που πιο αναλυτικά τεκμηριώνουν ή ισχυρίζονται ή θέτουν τα θέματα τα οποία προσπάθησα ε, γρήγορα να σας αναλύσω. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, και νομίζω ότι πρέπει σοβαρά να τα αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να τους απορρίψει αυτού του κανονισμού, πρέπει να απορρίψει τι προτάσει τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you um, ευχαριστώ πολύ. Να πεισαφηνήσω τώρα προς τα μέλη ότι θα προχωρήσουμε τώρα στις, ε, ε, στα σχόλια για την έκθεση της Ελίζα και μετά σκιώδες της και μετά θα κάνουμε τη διαδικασία catch the eye ε, όλων των μελών δηλαδή που θέλουν να μιλήσουν είτε για τη μία είτε για την άλλη έκθεση. Έχω 7 εγγεγραμμένους στη διαδικασία catch the eye. Ελίσσα για την έκθεσή σου. Ευχαριστώ λέει η Ελίζα. Μια στιγμή Ελίζα. Ο Βέρνερ θέλει να, να πει κάτι διαδικαστικά. Βέρνερ. Ναι, μέχρι, μέχρι τώρα μίλησαν δύο εκπρόσωποι των σκιωδών εισηγητών. Μα έτσι δεν θα γίνεται τίποτα, δεν, κάνουμε δουλειά. Εάν κάποιος δεν είναι παρόν, δεν είναι δυνατόν να, παρεμβαίνει και να από μια λίστα. Δεν είναι η διαδικασία αυτή. Νομίζω... Μέχρι στιγμής ε, είχα σκιώδη συγητέ που έλαβαν το λόγο και δίνω το λόγο στην ε, Ελίζα και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία η οφθαλμοσυλληπτική που είναι αυτό που ζήτησαν και οι συντονιστέ να είναι διαδικασία. Η Ελίζα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη κυρία Πρόεδρε. και θα ήθελα να ομαδοποιήσω τα προβλήματα σε τρεις μεγάλες ομάδες επί τη βάση των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Μια πρώτη ομάδα αφορά θέματα που πρέπει να υπόκειται σε μια πολιτική απόφαση και να προηγηθεί πολιτική συζήτηση και μέσα σε αυτά το θέμα μιας ενδεχόμενης συνένεση σε σχέση με το βαθμό ενσωμάτωσης ή μη της διακυβερνητικής συνθήκης. Εδώ έχουμε την πρόταση, την πρόταση αυτή που περιλαμβάνεται στην έκθεση Γκοζές και φαίνεται ότι καλύπτεται από μια γενική συνένεση και μπορούμε να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση και στις δύο εκθέσεις για το πολιτικό κομμάτι. Αλλά υπάρχουν πολλές τροπολογίες τώρα οι οποίες προσπαθούν να αλλάξουν ή να κάνουν ίσως πιο συγκεκριμένο και ασφαλές αυτό το οποίο προβλέπει η διακρατική συνθήκη και να το κάνουν και πιο συνεκτικό με όλα αυτά τα που έχουμε συζητήσει και εγκρίνει ως Κοινοβούλιο στην Εξάπτυχο. Επομένως, ό,τι ισχύσει για τη μία έκθεση θα ισχύσει για την άλλη και του κύριου Γκοζές και τη δική μου. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες προτάσεις τροπολογίας οι οποίες έχουν χαρακτήρα τροπο, ε, καινοτομίας, όπως η 210 των πρασίνων που ζητά να υπάρξει μια διαδικασία σε σχέση με τις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις, παράλληλα με αυτή που ακολουθείται για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από πολιτική άποψη, αλλά ανοίγει ένα τελείως διαφορετικό χώρο συζήτησης. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια πιο σε βάθος συζήτηση προτού αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια απόφαση απλώς ναι ή όχι. Μια τρίτη ομάδα που είναι πολύ σημαντική είναι αυτή που έχει να κάνει με το άρθρο 8 της πρότασης της Κομισιόν. Η Κομισιόν στο άρθρο αυτό ήθελε να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ αυστηρό καθεστώς για τις καταστάσεις αυτές που θεωρείται μια χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο να μην τηρήσει τα οφειλόμενα, τα υπεσχημένα ίσως. Αλλά αυτό για μας είναι μια ιδιαίτερα νεφελώδης έννοια. Δεν, μπο, μπορεί να υπάρχει μια τόσο αυστηρή διαδικασία και μια πρόσθετη πίεση προς τα κράτη-μέλη ότι η Κομισιόν δηλαδή μπορεί ξαφνικά να αποφασίσει ότι υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος, ένα κράτος να μην τα βγάλει πέρα, χωρίς να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο μπορεί να το ελέγξει κανείς και μετά θα απορρεύσουν πάρα πολλές συνέπειες για τη χώρα αυτή μετά από την απόφαση αυτής της Κομισιόν. Γι' αυτό το άρθρο 8 δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην πρόταση της Κομισιόν όταν υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος είναι τόσο άκαμπτος και τόσο ε, αυστηρός να επικαλείται λοιπόν απλώς τον κίνδυνο μιας χώρας να μην τηρήσει αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί η Κομισιόν για να εφαρμόσει ένα τέτοιο ε, δύσκολο και αυστηρό πλαίσιο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο οδηγεί εύκολα σε συνένεση. Υπάρχουν άλλα στοιχεία στα οποία έχουμε μια γενική συμφωνία. Παραγωγός χάρη να συναυθεί αυτή η διαδικασία με τη διαδικασία για το κρατικό χρέος. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι στις τροπολογίες τους. Εγώ είχα ήδη θέσει αυτό το ερώτημα του ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να φτιάνουμε αυτόνομους μηχανισμούς για την δημοσιονομική λιτότητα χωρίς συγχρόνως όπως πρότεινα εγώ να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το γενικό θέμα του κρατικού χρέους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε με ποιο τρόπο θα συναρμόσουμε όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ. Γιατί η πρόταση της Κομισιόν ήταν καταρχήν ενδιαφέρουσα, αλλά βλέπουμε ότι οι φιλελεύθεροι με την τροπολογία τους μιλάνε για ένα νομικό καθεστώς σε σχέση με το Ταμείο Απόσβεσης. Ορισμένοι λοιπόν θέλουν να προχωρήσουν με γοργά βήματα πάνω σε ζητήματα τα οποία είναι αμφιλεγόμενα και δύσκολα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο για να έχουμε μια διαδικασία η οποία θα γίνει δεκτή από όλους. Θα πάμε προς τα ευρωομόλογα, θα πάμε προς το Ταμείο Απόσβεσης και κάτω από ποιες συνθήκες και πώς θα μπορούσαμε εμείς να μπούμε σε λεπτομέρειες σε μια τέτοια λύση. ή θα σταθούμε στον κοινό παρανομαστή που είναι η εποπτεία του κρατικού χρέους και ο συντονισμός για τα θέματα του χρέους και αυτό το οποίο προτείνει ο Διογοφέο να υπάρχει κάποιο ταμείο έκτακτης ανάγκης σε σχέση με το κρατικό χρέος. Να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε κάποια αποτελεσματικά μέσα στη διαθεσή μας χωρίς να ανοίξουμε το κουτί της πανδώρας. Υπάρχει τώρα μια άλλη σειρά θεμάτων στα οποία μπορούμε νομίζω να είμαστε σύμφωνοι για το να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του Συμβουλίου Προϋπολογισμού και άλλων φορέων που καλούνται να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό αναφέρεται σε διάφορες τροπολογίες. Επίσης το να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο χρονοδιάγραμμα και όχι να δρούμε με πίεση χρόνου όπως αναφέρει κάπου η Κομισιόν στην πρότασή της. Υπάρχουν τροπολογίες εδώ διάφορες των φιλελευθέρων, της Μαριάν Τίσεν κτλ. Επίσης πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε και σε κάποια συμφωνία σε σχέση με την ιδέα του προγράμματο οικονομικής εταιρική σχέση μέσα στα πλαίσια όλης αυτής της διαδικασίας της πιο από κοντά παρακολούθησης του τι γίνεται σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και πάλι να επιτύχουμε μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει στο Six Pack, στην Εξάπτυχο και τις προτάσεις για το υπερβολικό ε, έλλειμμα και της αντανάκλασης στον προϋπολογισμό όλων αυτών των προτάσεων. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχάσουμε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει στο παρελθόν και να φτιάξουμε ασυνάρτητα νέα στοιχεία σε αυτό το νομοθέτημα. Ήθελα λοιπόν να ήμουν σύντομη και απλώς σας περιέγραψα ποιες είναι οι μορφές που έχουν οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ, Μαριάννου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για το έγγραφο το οποίο μας έδωσε και θα διευκολύνει πάρα πολύ την ε, συζήτησή μας γιατί είναι πάρα πολύ τεχνικά τα ζητήματα. Όσον αφορά το πρώτο σετ ερωτήσεων, ε, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια πολιτική συζήτηση. Το πρώτο θέμα αφορά το άρθρο 4 για το δημοσιονομικό σύμφωνο οπωσδήποτε το οποίο πρέπει να ενταχθεί. Έχω καταθέσει μια σειρά τροπολογίες ε, σχετικά και για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και για το λεγόμενο χρυσό κανόνα και τον αυτόματο ε, κανόνα διόρθωσης για το τι ακριβώς είναι ένας εξορροπημένος προϋπολογισμός ή ένας ε, προϋπολογισμός που αποκλίνει. Και αντιλαμβάνομαι πως οι συνάδελφοι δεν θέλουν να, ενταχθεί, να ενταχθούν οι λέξεις ε, αυτές ε, στον προπολογισμό. Θα τα δει η ομάδα μας και αν ε, μπορέσουμε να καταλήξουμε συμφωνία και σε άλλα λεπτά ζητήματα, νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε κάποια παραχώρηση σε αυτό και είμαι επίσης διατεθειμένη να αναζητήσουμε ένα κείμενο για το μισό της εκατό και το 1% μπορεί να φύγουν αυτά ίσως να μπουν σε ένα κείμενο το οποίο θα έχει συνταγματική φύση, αλλά να, το διατυπώσουμε διαφορετικά για να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με το σύμφωνο αυτό. Νομίζω λοιπόν πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο ναι θα λέει πράγματι ανεξάρτητη σε αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για να ελέγχουν εξ άντε και εξ αλλά πώς και με ποια βάση και νομίζω πως έτσι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία με όλες τις ε, ομάδες. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες ε, με αριθμούς για τους ε, προϋπολογισμούς σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός διορθώσεων. Τώρα, ο τρόπος, το εύρος και τα λοιπά μπορούν να έρθουν να ενσωματωθούν και νομίζω πως μπορούμε να παραπέμψουμε στους υφιστάμενους κανόνες από το εξαπλό πακέτο όπου γίνεται λόγος για διάφορους εθνικούς ε, κανόνες όσον αφορά τον προπολογισμό. Νομίζω πως ε, εάν τα λάβουμε αυτά υπόψη θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση κυρία Πρόεδρε. Για τους ανεξάρτητους φορείς μετά που θα κάνουν τις αξιολογήσεις στα κράτη-μέλη ε, βλέπω πως υπάρχουν αρκετές τροπολογίες, άλλοι θέλουν πράξεις κατεξοδότηση, άλλοι λένε να το κάνει η Κομισιόν. Εδώ πέρα αναρωτιέμαι κυρία εισηγήτρια, μήπως θα μπορούσαμε να εργαστούμε γρήγορότερα και να προβλέψουμε κάτι στον κανονισμό, να ζητήσουμε από την ε, Κομισιόν να ορίσει ποιες είναι οι απαιτήσει από ένα τέτοιο ανεξάρτητο όργανο. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε μια πράξη κατεξιοδότηση, γιατί να μην το κάνουμε τώρα, να υποβάλει τώρα προτάσεις η Κομισιόν και να μπει ήδη στον κανονισμό για να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. μην περιμένουμε μετά άλλον κανόνα να διαμορφωθεί. Είναι ήδη αρκετά περίπλοκα τα πράγματα. Αυτές οι προτάσεις ε, προς ε, την εισηγήτρια κατόπιν ε, στο άρθρο 5. Κυρία Πρόεδρε, Υπάρχει εδώ πέρα μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που θέλουν οι πράσινοι συνάδελφοι για παρακολούθηση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Ναι, συμφωνώ εδώ πέρα με την εισηγήτρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αλλαγή. Δεν είναι μια απλή ε, τροπολογία. Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και θα είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο ε, προτινόταν αρχικά. Οπότε ε, επί της αρχής θεωρώ πως πάει πάρα πολύ μακριά, αλλά επίσης πρέπει να δούμε ε, εάν βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο τα, τα πράγματα. Νομίζω πως ε, η, Ευρώπη, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 μιλάει εντάξει για ανάπτυξη και ε, θέσεις εργασίας και βεβαίως αναφέρεται στους προϋπολογισμούς, πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη κατόπιν ένα ερώτημα προς την εισηγήτρια για τη διαγραφή του άρθρου 8. Νομίζω πως είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η κυρία Φερέρα λέει πως δεν μπορεί να το στηρίξει γιατί δίνει πάρα πολλές αρμοδιότητες στην Κομισιόν. Διαβάζοντα αυτή την πρόταση όμω εδώ πέρα, ούτω ή άλλω ε, δίνουμε τη δυνατότητα στην Κομισιόν να κινηθεί αυτόνομα και να αποφασίσει μόνη τη. Αλλά ε, εμείς προτείνουμε η Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις ε, οι οποίες θα συζητηθούν με το Συμβούλιο ή καλύτερα με το Eurogroup έτσι ώστε οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη να ε, μπορέσουν να κρίνουν. Θα ήθελα να την υποβάλω αυτή την πρόταση στην κρίση της ε, εισηγήτριας και αν πρόκειται για περισσότερο από ένα κράτος μέλος αλλά για, για γενικότερες νομίζω πως μπορεί να γίνει η συζήτηση εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. Κατόπιν υπήρχαμε, υπήρχαν ερωτήματα της εισηγήτριας για το Εύρος, ε, άρθρο 2.3 και 3.3. Νομίζω πως είναι σημαντικό να υπάρχει μία διέξοδος κινδύνου. Εάν ε, δεν μπορέσει να καταλήξει σε υπολογισμό στο τέλος του έτους ένα κράτος μέλος, να υπάρχει μία δυνατότητα να κινηθούμε 12 τιμόρια κτλ. Βλέπω και άλλες ε, τροπολογίες στο να αντικαταστήσουν το κεντρική κυβέρνηση, το γενική κυβέρνηση με το κεντρική κυβέρνηση. Μπορούμε να το συζητήσουμε σε μία άτυπη συζήτηση. Αυτό είναι πρόβλημα όσον αφορά τα ομοσπονδιακά κράτη και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς ονομάζουμε τα πράγματα και το τι ζητάμε από τα κράτη-μέλη. Και μετά, κυρία Φερέρα, η άποψή μας για το άρθρο 5.3 σχέδια προϋπολογισμού και έκδοση χρέους. Όσον αφορά την έκθεση χρέους, ούτε υπέρ είμαστε, ούτε κατά. Νομίζω πως μπορούμε να το αφήσουμε όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύμφωνο. Δηλαδή όταν σκοπεύει να εκδώσει χρέος ένα κράτος μέλος να προειδοποιεί. Αλλά δεν μας φαίνεται κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει στο σχέδιο προπολογισμού ένα έτος πριν ή ενάμιση έτος πριν. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Οπότε ναι να υπάρχει μια παρακολούθηση αλλά να το αφήσουμε όπως υπάρχει στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο στην ε, διακυβερνητική συνθήκη και να μην ε, ε, συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο προπολογισμού που θα υποβάλλεται σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό κατόπιν άρθρο 6 για το χρονοδιάγραμμα και εμείς έχουμε υποβάλει ε, τροπολογίες η κυρία Φερέρα θέλει να γίνει πιο νωρίς η αρχή εμείς θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ νωρίς ειδικά αν δούμε τις οικονομικές προοπτικές οι οποίες γίνονται το φθινόπωρο, αλλιώς ε, θα βασίζεται το κράτος μέλος σε ξεπερασμένες ε, δημοσιονομικές ε, προβλέψεις. Οπότε, καλό είναι να παραμείνει η αρχή της διαδικασίας 15 Οκτωβρίου. Εάν η Κομισιόν θεωρεί πως πρέπει να αναθεωρηθεί κάτι, μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Εάν μετά είναι αναγκαίο να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να είναι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου έτσι ώστε να έχουν και τα εθνικά κοινοβούλια 6 εβδομάδες καιρό. Θα πρέπει να υπάρχει ε, εγκαίρος το σχέδιο στα εθνικά κοινοβούλια για να μπορούν και τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν την ε, αυτονομία τους και πρέπει να σεβαστούμε τα εθνικά κοινοβούλια και να έχουν 6 εβδομάδες στην ε, διάθεσή τους. Επίσης κάτι το οποίο βρίσκω σημαντικό κυρία Πρόεδρε, πως η Κομισιόν ε, λέμε πως θα πρέπει εδώ πέρα να μιλάει ε, μόνο όταν υπάρχει κάποιο ε, πρόβλημα μόνο. Εάν είναι εντάξει ο προπολογισμός δεν χρειάζεται να πει τίποτα η Κομισιόν, δεν χρειάζεται τώρα να πνιγούμε στην γραφειοκρατία. Τώρα, για το Ταμείο Διάσωση, θα σας δώσω την προσωπική μου άποψη. Δεν έχω τίποτα εναντίον. Είναι ένας από τους πιθανούς μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Αλλά τώρα να μπει εδώ μέσα χωρίς να έχουμε προτάσεις και συγκεκριμένα να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, δεν ξέρω, μου φαίνεται πως παραπάει. Δεν έχει σχέση με την παρακολούθηση. Αλλά όπως ε, λένε ούτως ή άλλως και αυτοί οι οποίοι κατέστησαν την πρόταση αφορά απλά το τεράστιο χρέος το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εδώ πέρα μιλάμε μόνο για παρακολούθηση. Και καλό είναι να μείνουμε στο θέμα μας. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν άλλοι 12 συνάδελφοι. Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Θα σταματήσω εδώ. Δεν είπα τίποτα για τον κύριο Γκοζές και ως σκιώδη ηγέτρια του ΕΛΚΑ πρέπει να απαντήσω τουλάχιστον σε ερωτήσεις ε, τη... της Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος, αλλά όλοι θέλουν να, να μιλήσουν. Και το KTI δεν βλέπω να το μέρα Ραμόν. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Τώρα ξεκινάμε τις ε, διαπραγματεύσεις ε, επί του εγγράφου. Πρώτον, ως φιλελευθεροί εμείς στηρίζουμε τις τροπολογίες, ε, οι οποίες ενισχύουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα σας καταπλήξω γιατί ούτως ή άλλω αυτή ήταν η γραμμή που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια η φιλελεύθερη ομάδα. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αυτή δεν είναι πολιτική κρίση. Μάλλον όχι, έκανα λάθος, ε, ε, λέει ο μιλητής. Δεν είναι μονάχα οικονομική η κρίση, είναι και, η πολιτική, είναι και πολιτική. Επομένως πρέπει να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες και την δύναμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί διαφορετικά ε, τα πράγματα θα συνεχίσουν όσοι έχουν και οι κυβερνήσεις θα φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Εάν συνεχίσουμε με αυτά που κάναμε τα τελευταία χρόνια, οπωσδήποτε ε, θα συνεχίσουν ε, οι δημαγωγικές κυβερνήσεις αυτές τις επικίνδυνες ε, συμπεριφορές. Θα πρέπει να δώσουμε επίσης η ενισχυμένη θέση της Επιτροπής σε σχέση με το Συμβούλιο και δεν μπορώ να κατάλαβω σε αυτόν τον κανονισμό και δεν καταλαβαίνω ακόμα αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν το Συμβούλιο να έχει μεγαλύτερη επιρροή ενώ έχει αποδειχθεί ότι στην ουσία είναι μια λέσχη φίλων ε, που ο ένας στηρίζει τον άλλο γιατί φοβούνται ότι θα του συμβεί αργότερα αυτό που συνέβη στους άλλους ε, ε, προηγούμενα. Επίσης στηρίζουμε όλες τις τροπολογίες οι οποίες ζητούν ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε περισσότερο διάλογο, θέλουμε περισσότερη πολιτική δημοκρατική λογοδοσία και κατά αυτή την έννοια έχω υποβάλει τροπολογία ε, ζητώντας μεγαλύτερη νομιμοποίηση για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κατά την άποψή μας να εκλέγεται και από τα μέλη του σώματος μεταξύ των μελών. Ε, that we uh, ε, και, και θέλουμε μεγαλύτερη νομιμοποίηση γιατί ο πρόεδρος Μπαρόσο τα τελευταία χρόνια ε, σε πολύ κρίσιμα σημεία της κρίσης ήταν εξεφανισμένος. Τρίτον, ως φιλελεύθεροι στηρίζουμε όλες τις τροπολογίες οι οποίες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα συμφωνήσουμε εδώ και με τους πράσινους, να δώσω κάποια παραδείγματα. Η διαφάνεια δε αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε ε, τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο στις ομόσπονδες χώρες. Ένα παράδειγμα. Χθες είχαμε εκλογές στην Ανταλουσία που είναι η μεγαλύτερη ε, ευρωπαϊκή περιφέρεια. Εκεί δεν υπάρχει ακόμα προϋπολογισμός από την εθνική κυβέρνηση γιατί είχαμε ε, ακριβώς αυτές τις εκλογές στην Ανταλουσία θα υπάρξουν και άλλες εκλογές ε, στην Ευρώπη, σε διάφορες περιοχές και επομένως και η Επιτροπή θα πρέπει εδώ να παίξει ρόλο υποπτίας ε, και στα, στους περιφερειακούς προϋπολογισμούς. Ε. Γιατί μια χώρα μπορεί να μην έχει προϋπολογισμό και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλη την Ευρωζώνη γιατί ας πούμε έγιναν εκλογές σε μια περιφέρεια, σε μια χώρα μέλος. Άλλο σημείο, όσον αφορά τώρα τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Εμείς ξέρουμε ότι ο ρόλος αυτός πρέπει και μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικός σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες στην ομάδα μου όσον αφορά την ε, αύξηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Ε, ζητώ λοιπόν να μάθω. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να μπλοκάρουν ε, κάποιες συμφωνίες. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις γνωμοδοτήσεις μας ή τις αποφάσεις μας γιατί αυτή είναι κόκκινη γραμμή για την Άλντε. Να υπενθυμίσω δε στους συναδέλφους ότι εάν θέλουν τα συνδικάτα να παίξουν όλο ε, στην διαδικασία α, ας πούμε ε, δημιουργίες ε, νομοθεσίας μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες ας πούμε. Επίσης, δύο σημεία. Πρώτον, να μην ε, ε, προχωρήσουμε σε ε, θεσμοθέτηση των πιστοτικών, των πιστοτικών Has no been one country default. στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχουμε ταυτόχρονα προετοιμαστεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση τους. Δεύτερον, πολύ με απασχολεί το θέμα ότι ε, ορισμένοι ιδιώτες επενδυτές ε, θα έχουν ε, μεγάλο τμήμα ομολόγων χρεών, κρατικών χρεών και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί δεν θα είναι πολλοί επενδυτές οι οποίοι μέσα από κουρέματα και τέτοιες διαδικασίες θα θέλουν πλέον να επενδύουν σε ορισμένες χώρες. Είναι γεγονός ότι ότι θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να υπάρξει ένα πολύ συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου καταστάσει και στο μέλλον. Ο Ντέρκ μίλησε, δεν θα ξαναμιλήσει. Φίλιπ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ίσως ε, να νομίσατε ότι ο προλαλής σας ε, ότι ο, ο, Σβέν μάλλον ότι προηγουμένως έκλεψε την ομιλία μου αλλά δεν τα κατάφερε τελείω. Θα κάνω λοιπόν μερικά σχόλια εδώ. Όταν λέτε ότι το Συμβούλιο είναι μια λέσχη φίλων, θα πρέπει να σας προειδοποιήσω για τις επιθέσεις κατά του Συμβουλίου. Ακούω πολλά τέτοια από τους φιλελεύθερους, <clears throat> αλλά έχουν εκλεγεί. Και μιλάω με ελευθερία γιατί δεν είναι πολύ πράσινη στο Συμβουλίο. Δεν πρέπει όμως να αρχίσουμε να κατηγορούμε και να περιφρονούμε αυτούς που είναι εκλεγμένοι όταν θέλουμε να έχουμε δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν μας αρέσει το αλογοπάζαρο που γίνεται στο Συμβούλιο. Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και πολύ περισσότερη από ό,τι η Κομισιόν από εκλογική έποψη. Δεν πρέπει λοιπόν να στρεφόμαστε κατά του Συμβουλίου. Παρά το γεγονό ότι είμαι φεδεραλιστή, το λέω αυτό. Μαριάν, τώρα, όταν λε ότι τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμιση είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ του, αυτό είναι το πρόβλημα κάποιος ο οποίος έχει βρεθεί σε μια κυβέρνηση ξέρει ότι είναι άλλη η πραγματική λιτότητα, είναι μια μεγάλη πειθαρχία και άλλη η πειθαρχία σε σχέση με τις επενδύσεις που συνδέεται με στόχους όπως η Ευρώπη 2020 που ο κόσμος το παίρνει στο ψηλό πολλές φορές. Γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη υποχρέωση ότι είναι πιο επιτακτικές αυτές οι δεσμεύσεις μας ώστε να αρχίσουν να εμπλέκονται και στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Και θέλω να υπενθυμίσω και τις συστάσεις που έχει κάνει η Κομισιόν σε σχέση με τους προϋπολογισμούς. Βλέπετε πολλές από τις ε, συστάσεις που πηγαίνουν στον τομέα του συνταξιοδοτικού τομέα, της εργασιακής πολιτικής κτλ. Λοιπόν, η Κομισιόν συνδέει επομένως αυτά τα πράγματα με τους προϋπολογισμούς. Αντί να το παραγνωρίσουμε αυτό, θα πρέπει να επιμείνουμε εμείς να μπορούμε να κάνουμε την απαραίτητη σύνδεση. Και ζητώ από την Κομισιόν να το λάβει αυτό υπόψη. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ασταθής η όλη αρχιτεκτονική του στόχου της Ευρώπης 2020. Θέλουμε να εδραιώσουμε καλύτερα αυτούς τους στόχους, να έχουν και νομική βάση, ώστε να υπάρχει κάποιο έδαφος επί του οποίου να οικοδομηθούν αυτοί οι στόχοι στην πραγματικότητα. Πρέπει όμως να παροτρύνουμε τα κρατημέλη να κάνουν τα απαραίτητα και να συνδέσουν αυτά που κάνουν με την Ευρώπη 2020. Αυτό που δεν θέλω είναι ότι όταν προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα του προϋπολογισμού, να παίρνουμε μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν εξυπηρετούν, αλλά τροχοπεδούν και τους στόχους της Ευρώπης 2020. Πείτε ότι έχουμε μια διαδικασία screening βάσει της Ευρώπη 2020 των εθνικών προπολογισμών. Να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που γίνεται σε επίπεδο προϋπολογισμού ουσιαστικά ευνοεί την επίτευξη των στόχων της Ευρώπη 2020. Τέλος λοιπόν, το θέμα τη δημοκρατική νομοποίησης είναι κομβικό, το έχω πει και στο παρελθόν πολλές φορές, ότι όταν ζητάμε από όλα τα στρώματα του πληθυσμού να κάνουν σημαντικές θητείες και όχι λίγους και άτυχους μέσα στον πληθυσμό, τότε πρέπει να έχουμε πραγματικά μια σημαντική νομιμοποίηση σε πολιτικό επίπεδο και για την ε, διακρατική συνθήκη το σύμφωνο αυτό δεν έχει καμία ευκαμψία. Οτιδήποτε πάει στραβά μπορεί να καταστρέψει αυτό το μηχανισμό. Παράδειγμα, όταν μιλάμε για τις τράπεζες μπορούμε να σκεφτούμε ότι θέλουμε να πάμε από μια κατάσταση α που είναι υγιής σε μια άλλη κατάσταση β που είναι υγιής επίσης, αλλά παίζει ρόλο και ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Αν δεν ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο, μπορούμε να μην φτάσουμε ποτέ στο β και μπορούμε να καταστρέψουμε την οικονομία μας στη διαδικασία. Λοιπόν, χρειάζεται μια μεγάλη ευκαμψία, είναι απαραίτητη. Το ίδιο ισχύει και για τις κυβερνήσεις. Άμα θέλουν να φύγουν από μια κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη σε μια κατάσταση που είναι βιώσιμη, χρειάζονται χρόνο αν δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγάλες καταστροφές και στην οικονομία και στην κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ευκαμψία όχι στους κανόνες, αλλά και στον τρόπο, όχι μόνο στους κανόνες, αλλά και στον τρόπο που εφαρμόζει η Κομισιόν τους κανόνες. Αν λοιπόν το δεχτείτε αυτό, υπάρχει δυνατότητα συνένεσης που να περιλαμβάνει τους πράσινους. Ποιος θα φανταζόταν ότι χρειάζεται τόση πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Ο Μιγκέλ Πόρτος είναι ο τελευταίος σκιώδης εισηγητής και μετά ακολουθεί μια οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία. Γιατί τονίζω ότι αυτοί που έχουν κάνει τροπολογίες πρέπει να μιλήσουν πρώτοι. Ο Μιγκέλ. Ευχαριστώ, Σάρον. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Εμείς καταθέσαμε μία τροπολογία για να επαναπέμψουμε στην Κομισιόν και τους δύο κανονισμούς, επομένως συνολικά η θέση μας είναι πάρα πολύ επικριτική σε σχέση με το περιεχόμενο των προτάσεων της Κομισιόν. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο έχουμε μια τόσο αρνητική και επικριτική στάση είναι το ότι ο κύριος στόχος των δύο κανονισμών, όπως και να το δούμε, είναι ουσιαστικά να ενσωματώσουν το πακέτο ε, συνεργασίας που προβλέπεται από τη νέα διακρατική συμφωνία. Όλα αυτά λοιπόν να τα βάλουν μέσα στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα φυσικά οι συζητήσεις που γίνονται δεν λένε διαφορετικά πράγματα. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει η Ελίζα Φερέιρα όταν αναφέρει την αντίθεσή της στο 8ο άρθρο της πρότασης του κανονισμού της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο κίνδυνο μη αποτελεσματικής εφαρμογής κάποιων μέτρων, το οποίο είναι κάτι απόλυτα σαφές. Και το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ασαφείς έννοιες, ώστε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε κράτη-μέλη, τα οποία ήδη υφίστανται ένα δρακόντιο καθεστώς βάσει της ε, οικονομικής, ε, διαδικασίας οικονομικού συντονισμού. Του του λεχθέντος, θα ήθελα να κάνω άλλη μία παρατήρηση σε σχέση με την πρόταση των πρασίνων στο, στην τροπολογία 209, όπου οι πράσινοι προτείνουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με επενδύσεις και απασχόληση στα εθνικά πρόγραμμα μεταρρύθμισης να αντιμετωπιστούν και να μην συμπεριλαμβάνονται, να εξαιρούνται όταν υπάρχει το θέμα της μη εφαρμογής κάποιων μέτρων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βρούμε και έναν τρόπο να πείσουμε τη Γερμανία να προχωρήσει σε μια οικονομική ανάπτυξη και αυτό το υποστηρίζω. Η ουσία της πρότασης αυτής είναι ότι όλο το πακέτο οικονομικού συντονισμού, όλο το σύστημα οικονομικού συντονισμού ουσιαστικά έχει να αντιμετωπίσει δύο αφεντάδες, και την ανάπτυξη και τη λιτότητα. Δεν επιλέγει σε στρατηγικό επίπεδο ποιος είναι ο στόχος αυτής της οικονομικής διαδικασίας, της διαδικασίας οικονομικού συντονισμού. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Είναι μια σχιζοφρένεια. Αυξάνεται ο μηχανισμός κυρώσεων στους οποίες βασίζεται το σύστημα του συντονισμού, χωρίς όμως να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των δυσκολιών που αντιμετωπίσουν κάποιες χώρες. Ζητά από την Πορτογαλία να επενδύσει όταν το συνολικό πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο ύφεση και όταν ακόμα και η ίδια η Κομισιόν εξακολουθεί να τονίσει ότι σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα υπεσχημένα δεν πρέπει να πάνε Διαρθωτική πόληση στην Πορτογαλία. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν λοιπόν. Τρίτη παρατήρηση. Σε σχέση με την κοινή διαχείριση του κρατικού χρέους και του Ταμείου Απόσβεσης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση και πρέπει να τη συζητήσουμε περισσότερο σε βάθος. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που εμπεριέχεται σε αυτή την ε, πρόταση είναι οι προϋποθέσεις για ένα ταμείο απόσβεσης γιατί είναι πραγματικά οι προϋποθέσεις υδρακόντιες των πολιτικών λιτότητος. Σημαίνει αυτό ότι τα επόμενα 20 χρόνια η Ελλάδα που έχει ένα δημόσιο χρέος 160% του ΑΕΠ θα πρέπει να κατέβει στο 60% του ΑΕΠ μειώνοντας το 1 20 του χρέου της κάθε χρόνο. Ποιος θα μου πει πώς, η Ελλάδα, πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει αυτή την προϋπόθεση την οποία θέτουν οι φιλελεύθεροι σε μια απαράγραπτη προϋπόθεση για να μπορέσει να υποφεληθεί από το Ταμείο Απόσβεσης. Ή μου πώς θα υπολογιστεί το διαρθρωτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα. Κανείς δεν μου έχει δώσει το μαθηματικό τύπο με τον οποίο υπολογίζει κανείς το διαρθρωτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα. Πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει ο οικονομικός κύκλος τι είναι υπερκυκλικό, τι είναι αντικυκλικό. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ προβληματικά για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα διαβάσω, είναι αναομάδες, ε, το ποιο θα μιλήσω. Astrid Lulling, Werner Langen, Roberto Galtieri, Liam Sanchez and myself, though I guess I'll slip off the end. Uh, και εγώ, αν και μάλλον στο τέλος δεν θα μιλήσω. Γκίνερ, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα νομίζω πως είναι σημαντικό το χρηματοοικονομικό συμβούλιο να είναι πλήρω ε, ανεξάρτητο. Και αυτό ισχύει για τα πάντα, στατιστικά στοιχεία κτλ. Αν δεν μπορούμε να το εγκινηθούμε αυτό, θα μπούμε στην ίδια διαδικασία που είχαμε και την τελευταία φορά που συζητήσαμε αυτό το θέμα. Θα έχουμε ηθικές κρίσεις παρά κανόνες. Και όταν μιλάμε για ευελιξία, υπάρχουν δύο σκοπιές στην ευελιξία. Είτε μπορούμε να έχουμε ευελιξία στην εισαγωγή των πολιτικών ή στην ερμηνεία των κανόνων και δεν θέλω να έχουμε ευελιξία στην ερμηνεία των κανόνων γιατί ακριβώς αυτό είχε συμβεί με το παλαιό σύμφωνο σταθερότητα. Ερμηνεύονταν με διαφορετικούς τρόπους και δεν είχε αξία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι για κάποια πράγματα ότι θα έχουμε κανόνες και όχι την κρίση των πολιτικών και ανησυχώ λίγο για κάποια κομμάτια της ε, έκθεσης ε, της ε, κυρίας Φερέιρα γιατί εδώ πέρα υπάρχει περιθώριο για κρίση και όχι για αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και πρέπει να το τονίσουμε αυτό πολύ περισσότερο γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και αναφέρομαι σε κάποιες παρεμβάσεις δεν είναι πως έχουμε λίγα κίνητρα για την οικονομία, γιατί αν δούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια ή ακόμα και την ιστορία του Συμφώνου Σταθερότητας, είχαμε πάρα πολλά ελλείμματα για να δοθούν κίνητρα στην οικονομία. Και το πρόβλημα είναι πως δεν λειτουργεί αυτό και πολλές κυβερνήσεις ε, χρησιμοποίησαν αυτές τις ευκαιρίες για να αποφύγουν τις διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Όσο πιο ε, αυστηρούς κανόνες, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από την κρίση και θα έχουμε και ευκαιρίες ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω την ε, ανάγκη στο μέλλον να τηρούμε κανόνες, ε, να τηρούμε αυστηρά κανόνες σαφείς και ε, εύκολους. Ρομπέρτο. Ευχαριστώ. Δύο σημεία θα αναφέρω μόνο, στα οποία αναφέρονται και οι τροπολογίες μου. Πρώτα απ' όλα, δημοκρατική λογοδοσία. Συμφωνώ με τον Ζαπολ ότι η πρόταση της Επιτροπής αφήνει μόνο στην Επιτροπή ε, την ευθύνη για πολύ σοβαρές αποφάσεις, ε, υπερβολικά σοβαρές για να μην έχουν ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση. Όμως από νομικής απόψεως δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η νομιμοποίηση θα πρέπει αποκλειστικά να προέρχεται από το Συμβούλιο. Προσωπικά πιστεύω ότι μια και πρόκειται για μια εποπτεία και που επομένως αφορά ε, τη νομική βάση του άρθρου 121, όπου το 121.6 αναφέρεται στη συναπόφαση, δεν καταλαβαίνω γιατί ε, δεν μπορούμε να ε, δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν μεγαλύτερο ρόλο, τον οποίο εγώ προβλέπω ακριβώς στις τροπολογίες μου και με διαφορετική μορφή ανάλογα με το είδος παρέμβασης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική πίεση και σκόπιμο θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατελάχιστον να ε, ζητήσει όσο γίνεται μεγαλύτερο ρόλο τουλάχιστον ε, όποιον ε, νομίμως και βάσει των νομοθετικών πλαισίων μπορεί να ζητήσει. Δεύτερον, Fiscal Compact. Έχω και εδώ νομικές έτσι, αμφιβολίες όσον αφορά την ε, δυνατότητα αναφοράς στο Fiscal Compact ε, σαν ε, πρόσθεση του τροποποιημένου 1466 η μόνη μορφή θα μπορούσε κατά την άποψή μου ε, να είναι να ενσωματωθεί τροπολογία ε, στον κανονισμό 1466 γιατί θα είχαμε δύο διαφορετικούς κανονισμούς που αφορούν το ίδιο ε, θέμα. Αυτό είναι ουσιαστικό σημείο, δεν είναι δικολαβίστικο. Ε, γιατί κατά την άποψή μου το, ε, ο λόγος για τον οποίο είναι δόκιμο να ενσωματωθούν ε, de facto τα στοιχεία που αναφέρονται και προβλέπονται στο Fiscal Compact και να ενσωματωθούν λέω στο Σύμφωνο Ανάπτυξης βασίζεται στο γεγονός ότι στο Fiscal Compact ζητείται να ενσωματωθεί, να εγγραφεί στις ε, εθνικές ε, διατάξεις το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να έχει πάντα τον πρωταρχικό ρόλο και τη δυνατότητα τελικού ελέγχου έτσι όπως αυτός αναφέρεται στα, στις ιδρυτικές συνθήκες και στην συνθήκη λειτουργίας. Και επομένως ε, ε, στον κανονισμό 1466-67 τροποποιημένο από το Six Pack θα πρέπει να ε, υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση της διορθωτικής ισορροπίας structural balance βάσει βάσει όλων των ε, αρχών που διέπουν αυτήν την structural balance. Από πολιτικής απόψεως νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στο μέλλον, στους επόμενους μήνες δηλαδή, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κοινό έδαφος ε, έτσι ώστε να μας επιτρέψει να ε, έχουμε παράλληλα και δημοσιονομική πειθαρχία αλλά και μέτρα για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να συγχαρώ τους δύο εισηγητές γιατί έχουν καταφέρει στο, στα έγγραφά τους να παρουσιάσουν θέσεις και κατευθύνσεις που μπορούν να αριστούν μια συνένεση και επίσης γιατί έχουν προσπαθήσει να συνδέσουν όλα αυτά με το six-pack, την εξάπτυχο και με τον τρόπο αυτό μπορούν να διευκολύνουν την ταχεία λήψη απόφασης για τα θέματα αυτά. Εμείς σαν πολιτικοί πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας ότι οι πολίτες περιμένουν από εμά να υπάρξει μια ταχεία λύση και απόφαση και θα πρέπει να γίνει σαφής πολύ σύντομα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Έχω πέντε σημεία τα οποία θέλω να θίξω σε σχέση με το σύνολο των τροπολογιών που έχω καταθέσει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα της συνεκτικότητος αυτού, αυτών των δύο κανονισμών και του six-pack. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια συνέχεια μεταξύ των δύο. Παραδείγματα. Ο οικονομικός διάλογος. Δεύτερον, η αντίστροφη πλειοψηφία σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων της Κομισιόν. Δεύτερον, η διαχείριση του χρέους με ολοκληρωμένο τρόπο και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα προσοχή σε ορισμένα θέματα. Θα πρέπει όλες οι αποφάσεις να περιλαμβάνουν και κάποια επιφύλαξη, διότι αν γίνονται να μην, γίνονται, δημοσιεύονται αυτές οι απόφασεις, γιατί θα έχουν επιπτώσεις στην αγορά. Τρίτον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξή. Ότι θα πρέπει να διαλευκανθεί αν χρειάζεται ή όχι μία αλλαγή των συνθήκων. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις ακόμα και μέσα στην ε, ίδια την Κομισιόν για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά ταμεία, το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, ότι πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη και πέμπτο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί για τον προϋπολογισμό. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα ίσον θέμα, αλλά μπορεί να μας οδηγήσει σε πρακτικά προβλήματα εφαρμογής τους κανονισμούς και επομένως να θίξει το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Γι' αυτό κατέθεσα σε σχέση με τις ημερομηνίες που προβλέπονται στις προτάσεις αυτές. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Jean Paul για το γεγονός ότι έχει αφαιρέσει ένα τμήμα της τροπολογίας που προέτεινε να απεληθεί ο χρυσούς κανόνας της ε, διακυβερνητικής συμφωνίας. Έτσι λοιπόν δεν ήταν άχρηστη η μπλε κάρτα που του σήκωσα στην Ολομέλεια και σε σχέση με αυτό δεν είναι άψογη η Κομισιόν λόγω της, ε, διαδικασίας, λόγω της διατύπωσης που έχει σε κάποια ε, στοιχεία της πρότασής της. Δεν μπορεί ο χρυσούς κανόνας να εμφανιστεί στο παράγωγο δίκαιο γιατί όλα αυτά είναι αντίθετα με το άρθρο 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αν δεν υπάρξει λοιπόν μια τροποποίηση αυτού του άρθρου, δεν μπορούμε να εισαγάγουμε στο παράγωγο δίκαιο τον χρυσούν κανόνα. Θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι συνάδελφοι του ΕΛΚ, γιατί άκουσα κάποια ανησυχητικά πράγματα από τα χείλη τους και ίσως δεν έχουν συζητήσει απόλυτα με τον εισηγητή τους και τον συντονιστή τους. Εγώ έχω κάνει μερικές τροπολογίες μαζί με την Ελίζα για να εισαγάγουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στην έκθεση αυτή όταν αυτό είναι απαραίτητο. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, είμαι πολύ σκεπτικιστής σε σχέση με τα redemption bonds και το Ταμείο απο, Απόσβεσης. Μπορούμε να χρηματοδοτούμε λοιπόν για την ανάπτυξη σε μια χώρα που τη ζητάμε συγχρονώ να πάρει μέτρα τα οποία σκοτώνουν αυτή την ανάπτυξη και το κεφάλαιο 11, η ρύθμιση αντίστοιχη του κεφαλαίου 11 στι ΗΠΑ που ανέφερε ο Ζαν Πολ Γκοζέ, πολλοί θεωρούν ότι αυτό μπορεί να έχει αντικικό αντίκτυπο στα επιτόκια. Η πιο πραγματιστική και πιο απλή ε, λύση θα ήταν να έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο σταθερότητα μια άδεια να λειτουργεί σαν τράπεζα και έτσι να μπορεί να είναι καταπιστευματοδόχος του κρατικού χρέους, αλλά όλα αυτά τα θέματα απαιτούν μια αντιμετώπιση η οποία θα είναι πιο πραγματιστική. Ευχαριστώ. Η Αστρίδα. Πάρα πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε για μέσα από τις τροπολογίες μου. Στην έκθεση Γκοζέσα θέλω να υπογραμμίσω ότι έχουν σαν στόχο να συμμετέχει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή προγραμμάτων προσαρμογής στα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δεν το κάνω από κορπορατιστικό πνεύμα επειδή είμαι ευρωβουλευτής αλλά διότι θεωρώ ότι υπάρχει προσθέμενη αξία, σημαντική προσθέμενη αξία από τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τη δημόσια συζήτηση και θα υπάρξει πραγματικά ένα πλεονέκτημα να γίνονται δημόσιες συζητήσεις για τα προγράμματα αυτά προσαρμογής και με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί και μια μεγαλύτερη νομιμοποίησή τους για την Ελλάδα τώρα. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν θα πρέπει να τα δούμε σαν παράδειγμα και να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από αυτά. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία με αφήνουν εμβρόντιτοι. Δόθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία δόθηκαν για να βοηθηθεί η Ελλάδα ενώ από την άλλη πλευρά έχουν δαιμονοποιηθεί όλα αυτά τα ε, σχέδια ανάκαμψης τα οποία ουσιαστικά επιβάλλουν θυσίες και δάκρυα στον πληθυσμό της Ελλάδος. Αυτό μας δείχνει ότι οι προσπάθειες εξυγίανσης και βιωσιμότητας αν δεν έχουν παράλληλα την απαραίτητη διαφάνεια ουσιαστικά αποδυναμώνουν όλη αυτή τη διαδικασία και υποσκάπτουν αυτά τα οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά δεν έχει την δυνατότητα να παρέμβει 100% σε αυτή τη διαδικασία αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση του Κοινοβουλίου, να έχει το Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εκδίδει μια γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά, ιδίως όταν πρόκειται για την εφαρμογή προγραμμάτων λιτότητος, προσαρμογής και υπάρχει και μια προϋπόθεση για μια τέτοια γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορεί να έχει μια ταχεία απάντηση και όχι με τις διαδικασίες αυτές να περιπλέξει και να καθυστερήσει τη διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν δυνατότητα ταχείας αντίδρασης. Για να συμμετέχει το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των διακυβευόμενων και τουλάχιστον να βρει έναν τρόπο να επιταχύνει τις μεθόδους εργασίας του το Κοινοβούλιο. Γιατί αυτό το οποίο έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευίωνο. Υπάρχουν κανονισμοί που έχουν υποβληθεί από την Κομισιόν τον Νοέμβριο, το ΕΚΟΦΗΝ έχει ήδη συμφωνήσει τον Φεβρουάριο, όπως είπε και ο εισηγητής ο Ζωάν Πολ προηγουμένως, στην εισαγωγική του ομιλία, αλλά το Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα. Και κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και το κατεπήγον, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα παραγωγικό κάτι τέτοιο και επικοδομητικό. Κάθε άλλο. Βλέπω ότι κάποια από τα μέλη της Επιτροπής μας, ιδίως προς τα αριστερά, έχουν την, ε, τον πειρασμό να αφήσουν τα πράγματα να τρέχουν και να τα καθυστερούν. Εγώ τους ε, τους παρακαλώ να μην μπουν στον πειρασμό αυτό που μας οδηγεί σε μια παγίδα. Τα φάρμακα πρέπει να τα παίρνει κανείς στην κατάλληλη στιγμή και όχι να τα καθυστερεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική λύση για την εδραίωση των δημοσίων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαδικασία προσαρμογής, μια ευφυής διαδικασία ε, εφαρμογής για να αποφύγουμε την ύφεση που δημιουργούν. Αυτή είναι η άποψη μου λοιπόν. Ελπίζω ότι θα γίνει κατανοητό αυτό το οποίο αναφέρω και τα έχω συμπεριλάβει στις τροπολογίες μου και ζητώ και πάλι να μην καθυστερείτε τα πράγματα και τη λήψη αποφάσεως. Ο Αντολίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι τροπολογίες που έχω παρουσιάσει στην έκθεση Γκοζές, αυτό το οποίο επιζητούν, είναι να συμβάλλουν στην προσπάθεια του εισηγητή να βελτιώσει την πρόταση της Κομισιόν και να δώσει και πρόσθετο υλικό για να μπορέσουμε να έχουμε ε, συζήτηση και διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ουσιαστικά μιλάμε τώρα για την οικονομική διακυβέρνηση μέσα στην ζώνη του ευρώ και το πώς αντιμετωπίζονται οι χώρες που έχουν οικονομικά προβλήματα. Κατά την άποψή μου λοιπόν, η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να ε, εμπλουτιστεί με τέσσερις ιδέες που να είναι σαφείς. Πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη, πιο δίκαια, πιο αποτελεσματική και πιο νομιμοποιημένη. Το πρώτο σημαίνει πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία των χωρών που έχουν προβλήματα. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η διαδικασία ενισχυμένης εποπτείας σημαίνει και ενισχυμένη συνεργασία και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η φιλοσοφία που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε. Δεύτερο, θα πρέπει να είναι πιο δίκαια η εφαρμογή αυτών των μέτρων. Αυτό το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να ξαναφέρουμε μια χώρα στην τροχιά της βιωσιμότητας. Συμφωνώ. Αυτή η βιωσιμότητα όμως του κρατικού χρέους θα πρέπει να έχει και μια παράμετρο αναφοράς μέσα στην ίδια την ζώνη του ευρώ. Δηλαδή να απαιτείται μια προσπάθεια από τη χώρα αυτή η οποία να είναι αφεαυτής η προσπάθεια αυτή βιώσιμη και όχι υπερβολική. Όταν μιλάμε τρίτον για την αποτελεσματικότητα, σχέδιο προσαρμογής θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα συνοδευτικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει οικονομικά και νομισματικά μέτρα παραδείγματος χάρη να διατηρήσουμε την ε, λειτουργία των πιστοτικών ιδρυμάτων να καπατάξουμε τη φοροδιαφυγή να εμποδίσουμε τη φυγή των κεφαλαίων να τηρήσουμε λοιπόν μία σειρά από στόχου, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της ανισορροπίας μέσα στο κράτος μέλος αυτό. Και εδώ χρειάζεται συνεργασία των άλλων χωρών. Και το τελευταίο στοιχείο είναι η νομιμοποίηση. Δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι είναι οι πιστωτές οι οποίοι επιβάλλουν στις χώρες αυτές κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να επιμείνουμε στην λογική την ενωσιακή και στη λογική την κοινοβουλευτική. Μου φαίνεται ότι ο κ. Κόζες λέει εντάξει το Συμβούλιο έχει μια ευθύνη για τα θέματα. Φυσικά έχει μια ευθύνη αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό η πρότασή μου αυτή τη στιγμή θα ήταν πάρα πολύ σαφής. Δηλαδή τα σχέδια σταθεροποίησης και τα συνοδευτικά σχέδια να εγκρίνονται με τη διαδικασία των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό θα δώσει και στο Κοινοβούλιο να έχει κάποιο λόγο στα θέματα αυτά και η φόρμουλα αυτή των κατεξουσιοδότηση πράξεων έχουν μια γενική κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να ανταποκρίνονται και σε αυτά που θέλει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Βέρνερ. Ναι. κάτι με αυτή τη συζήτηση. Έχουμε το εξαπλό αυτό πακέτο το οποίο το εγκρίναμε με πολιτική πλειοψηφία. Εντάξει, κάποια μέρη ήταν επίμαχα. Οι διευκρινήσεις ε, της ε, Κομισιόν ήταν κάτι το οποίο ήθελε εδώ πέρα η πλειοψηφία και διαπιστώνω τώρα πως ε, αυτό το οποίο προτείνει ο Ζαν Πολ Γκοσές μετά από αυτές τις ξεκάθαρες πολιτικές τοποθετήσεις αμφισβητείται όπως ε, και από τη συνάδελφο Φερέρα, αμφισβητείται ε, το πόσο ε, θα υπάρξει σοβαρότερη υποπτία. Εμείς ζήτησαμε αντεστραμμένη ειδική πλειοψηφία για τις κυρώσεις και είχαμε ασκήσει κριτική στους Μέρκελ και Σαρκοζή για την συμφωνία της Ντοβίλ και μετά ε, καταφέραμε να περάσουμε το αντίθετο που ήθελαν ε, αυτοί οι δύο σημαντικοί ηγέτες και τώρα περνάμε το ε, αντίθετο. Δηλαδή τι θα γίνει, θα τα ξαναντιστρέψουμε όλα, απλά αναρωτιέμαι. Βλέποντας τα άρθρα 35 έως 38 τις τροπολογίες. Πάλι εδώ πέρα τι ζητάμε διατάξεις για να γίνει για να προξενήσουμε ουσιαστικά έναν ε, πόλεμο. Και αυτά τα οποία έχουμε εδώ πέρα ε, προβλέπονται στα άρθρα της συνθήκης. Το άρθρο 125 παραδείγματο χάρη ε, για ένα, σύμφω... για ένα ταμείο σταθερότητας κτλ. Αν παραδείγματο χάρη η κυρία Γκουγιάρ των Φιλελευθέρων θέλει να περάσει εδώ πέρα τα αγαπημένα της ε, θέματα. Δεν κολλάνε αυτά με το θέμα της έκθεσης και η κατηγορία των κομμουνιστών ότι α ναι ε, να απορρίψουμε τον κανονισμό αλλά μετά να λέμε πως ε, υπάρχει εδώ πέρα το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Όχι, αυτά είναι από τις 23 Νοεμβρίου 2011. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο πέρασε Δεκέμβριο. Οπότε έγιναν αυτές οι προτάσεις από την Κομισιόν προ συμφώνου με βάση την συζήτηση που ζήτησε δύο χρόνια, μετά από δύο χρόνια συζήτησης το Κοινοβούλιο με ευρύτατη πλειοψηφία. Και προσπαθούμε πάλι ξανά να τα εξασθενήσουμε αυτά τα πράγματα. Και πάμε δηλαδή σε, σε λάθος δρόμο αν θέλουμε πρώτον να αποδυναμώσουμε τους οργανισμούς αυτούς. Δεύτερον να λέμε πως δεν είναι δημοκρατικό όταν εμείς στην διαδικασία της συναπόφασης αποφασίζουμε. Και η τελευταία μου παρατήρηση για το χρονοδιάγραμμα. Η παρελκυστική αυτή τακτική να τα πάμε το φθινόπωρο. Όχι, λάθος. Επειδή αντιδράσαμε τόσο αργά ως πολιτικοί επιδεινώθηκαν τα προβλήματα και είναι τελείως λάθος να μην εργαστούμε τώρα γρήγορα. Για κάθε, για κάθε βλακεία τα πάμε γρήγορα. Κάνουμε γρήγορη διαδικασία και εδώ πέρα που θέλουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό ο οποίος θα αποτελέσει και βάση για ανάπτυξη, το αναβάλουμε γιατί κάποιοι συγητέ και σχεδόν συγητέ ε, δεν του άρεσε. Ε, αυτά είναι ανεύθυνα πράγματα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα κάνω μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Πολύ ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΩΣΑ ότι είναι πιο οικονομικά αποδοτικό να πάρει κανείς πιο δραστικά μέτρα και νομίζω ότι αυτή η πρόταση του Ζαν Πολ Γκοζέσε για σύστημα πτώχευσης τύπου άρθρου 11 ε, είναι, ε, πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή όντως θα πρέπει να δρούμε έγκαιρα, πρώιμα ε, γρήγορα. Και εγώ έχω υποβάλει ε, μια τροπολογία κατά αυτήν την έννοια και θα πρέπει να, αντιμετωπίσουμε τις αγορές ε, προ, έγκαιρα και να, τις, παίρνουμε και αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα τις εκπλήξουν, δεν θα τους δώσουν πάρα πολύ χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Εάν οι εισηγητές μπορούν να κάνουν πάρα πολύ σύντομες ε, παρεμβάσεις ε, να το κάνουν, αλλά πάντως θα πρέπει φαντάζομαι να μιλήσετε και διμερός και να δώσετε διμερός απαντήσεις. Ε, ο κύριος Γκοζές, πρέπει να πω ότι πραγματικά κάνω τα πάντα έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα και αυτό το λέω για να ε, μην ανησυχεί ο Βέρνερ. Να προχωράμε γρήγορα για να ψηφίσουμε στις 14 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Τα έχω ήδη ε, σημειώσει, έχω δει και τις ε, τροπολογίες αλλά έχουμε μπροστά μας και πολλές ακόμα συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές και επομένως σε εδώ έφετο χρόνο θα προχωρήσουμε έτσι ώστε η αξιοπιστία του κοινωνικού Κοινοβουλίου να μην υποφέρει. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο αυτούς που κατέθεσαν ε, τι τροπολογίε, αλλά και όλους αυτούς που συμμετέσχαν στη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ ευχαριστώ. Θα συζητήσω προσωπικά και διμερώς όλα αυτά τα θέματα, αν έχετε κάποιες ε, απορίες ή κάποιες αμφιβολίες που θα πρέπει να τις διαλευκάνω και να προσπαθήσω να καταλάβω και εγώ καλύτερα τη λογική τις επιχειρηματολογίες των τροπολογιών σας. Γι' αυτό πάλι και θέλω σας και πάλι να σας ευχαριστήσω για το θετικό πνεύμα με το οποίο γίνεται η συζήτηση. Ξέρουμε όλοι ότι όλα αυτά τα θέματα είναι τεράστια σημασίας και ότι οι δύο αυτές εκθέσεις είναι συμπληρωματικές με αυτά τα οποία αποφασίσαμε πριν από ορισμένου μήνες είναι δύσκολο να προχωρούμε με τέτοια ταχύτητα στην εκπόνηση νομοθεσία χωρί να προκύψουν ασυναρτησίε, τι οποίε φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφύγει. Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξουμε σε ένα κοινό εδρεωμένο κείμενο το οποίο μπορούμε να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ, Λέκη Πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε βεβαίω ε, το χρονοδιάγραμμα, αλλά η ψήφιση στην Επιτροπή θα γίνει η 25 ή 26 Απριλίου και σα προειδοποιώ πως ε, θα συνεδριάσουμε τότε Τετάρτη Πέμπτη και η 26η είναι Πέμπτη. Προσπαθούμε να δούμε πως η ψηφοφορία γίνει Τετάρτη ε, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε και σκοπεύουμε να πάμε ολομέλεια Ιούνιο ή Ιούλιο αναλόγως. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας. Ξεπεράσαμε το χρόνο αλλά είναι σημαντικό το θέμα. Περνάμε τώρα γρήγορα στο σημείο 6 η έκθεση της Άννης Ποδηματά για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και εξέταση τροπολογιών. Άννη. Ευχαριστώ Σάρων. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και ειδικά τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, που κατέθεσαν ε, τροπολογίες. Είμαι σίγουρη πως θα έχουμε ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συζήτηση και αναμένω τις συζητήσεις που θα συνεχιστούν με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Να υπενθυμίσω πως πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τρεις λόγους. Πρώτο πόλεμο για νέους πόρους, δεύτερον για να ε, διορθωθεί η υποφορολόγηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τρίτον για να αντιμετωπίσουμε τις ε, κερδοσκοπικές ε, βραχυπρόθεσμες τάσεις. Θεωρώ πως πρέπει λοιπόν να έχουμε τώρα μια συνεκτική προσέγγιση και να είμαστε σοβαροί όταν λέμε πόσο ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να υπηρετεί την πραγματική οικονομία. Νομίζω συνολικά πως ε, πρέπει τώρα να δώσουμε ουσία σε αυτά τα οποία λέμε. Δεύτερον, η επιτυχία του φόρου αυτού εξαρτάται βασικά από το πώς θα σχεδιαστεί που δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώριο φόρο αποφυγής. Δηλαδή θα πρέπει να ισχύει για το ευρύτερο δυνατό φάσμα προϊόντων και για όλα τα μέρη μιας συναλλαγής. Και θεωρώ πως υπάρχει αρκετός κοινό τόπος ε, υπ' αυτή την έννοια. Οπότε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη δικασία αυτή κατά την άποψή μου είναι να συμπληρώσει και να βελτιώσει την πρόταση της Κομισιόν για να ενθαρρύνει μια συμβιβαστική λύση στο Συμβούλιο. Να περάσω τώρα στις ε, τροπολογίες. Εάν αποκλείσουμε τις τροπολογίες που ζητάνε απόρριψη της πρότασης, οι υπόλοιπε ε, συνοψίζονται σε έξι κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα κάποιες τροπολογίες που προτείνουν εναλλακτικέ προς το φόρο αυτόν, όπως έναν ΦΠΑ ή κάποιον άλλο φόρο. Και πάλι νομίζω πως εδώ πέρα έχουμε ζήτημα συνέπειας, δεν θα πρέπει να προσφύγουμε σε εναλλακτικά μέσα φορολογίας, σε αυτό εδώ το κείμενο. Το να πάμε σε ΦΠΑ ή άλλους φόρους στο χρηματοπιστωτικό τομέα, θεωρώ πως δεδομένων των συνθήκων είναι ένας τρόπος να αποφύγουμε την συζήτηση και δεν θα πρέπει να είμαστε εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αυτοί που θα ξεκινήσουν μια τέτοια συζήτηση. Δεύτερον, επέκταση των usage και των AIF. Ήθελα σύντομα να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στο ζήτημα των συνταξιοδοτικών ταμείων γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Απασχολεί πολλούς συναδέλφους. τα ταμεία αυτά. Νομίζω πως αυτή είναι η πρόθεση της έκθεσης της Κομισιόν με την οποία συμφωνώ πλήρως. Ε, τα συνταξιδοτικά ταμεία θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συντηρητική επενδυτική στρατηγική μια στρατηγική δηλαδή η οποία είναι διακράτησης των χρεογράφων. Δεν έχουν στόχο την κερδοσκοπία. Με στόχο σύμφωνα δηλαδή με το στόχο του συνταξιωτικού ταμείου να πληρώσει δηλαδή μετά από 30 χρόνια μια σύνταξη. Όσον αφορά λοιπόν το... την επίδραση του φόρου αυτού στην απόδοση είναι αν υπάρχει στην τάξη του δεκαδικού ψηφίου και σύμφωνα με το σενάριο της Κομισιόν το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην αναθεωρημένη μελέτη αντικτύπου, ένα συνταξιοδοτικό ταμείο το οποίο ε, αντιπροσωπεύει 20 χρόνια αποταμιεύσεων από επίδοξους ε, συνταξιούχους θα είναι σαν να μην έδινε 100 ευρώ το μήνα ο επίδοξος συνταξιούχος, αλλά 99,995, μιλάμε δηλαδή για 0,005 Κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου είναι πως οι πρωτογενείς αγορές και οι συναλλαγές σε ακίνητα εξαιρούνται. Οπότε δεν θεωρώ πως υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα για ειδική μεταχείριση των συνταξιδοτικών ταμείων, εκτός εάν θέλουμε να τα ενθαρρύνουμε να ακολουθήσουν επικίνδυνες στρατηγικές, οι οποίες όπως έδειξε η κρίση μπορεί να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα στους ε, συνταξιούχους και τους πολίτες γενικώ. Uh, Αυτό το οποίο αξίζει να εξετάσουμε ως ιδέα είναι να υπάρξει μία δυνατότητα επιστροφής χρημάτων όπου οι επενδυτές λιανικής οι οποίοι αμέσως ή εμέσως μέσω επενδυτικών ε, οχημάτων ε, υπόκεινται σε αυτό το φόρο να λαμβάνουν πίσω τα χρήματά τους υπό ε, την προϋπόθεση ότι θα είναι τα ποσά κάτω από ένα ορισμένο ποσό ή πως θα ισχύει ο φόρος για κάποια ε, ποσά και πάνω. Αυτά ως μια προσπάθεια αναζήτησης ε, συμβιβασμού. τρίτων τροπολογίες για ενίσχυση τη νομική βάσης για να έχουμε μια ενισχυμένη συνεργασία. Στηρίζω τις ε, τροπολογίες, αλλά θεωρώ πως θα πρέπει να μπουν στα εκτιμώντα για να σεβαστούμε την διαδικασία. Τροπολογίες κατόπιν που ε, σχετίζονται με το ύψος Θεωρώ πως η πρόταση της Κομισιόν για, για μια ελάχιστη εναρμόνιση του ύψους είναι η σωστή. Ε, είναι αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή για το ΦΠΑ, έχει αποδειχθεί μια επιτυχημένη προσέγγιση και είναι η σωστή προσέγγιση όσον αφορά και τον φόρο αυτόν. Όσον αφορά το ύψος, λοιπόν, θα προτιμούσα να παραμείνει σε μια αρχική φάση χαμηλό, και η ε, ομάδα ειδικών του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όπως πρότεινε η συνάδελφη Κάνφερ και Γκίγκολτ να έχει την εντολή να επανεξετάσει την κατάσταση και να προτείνει τροπολογίες και αλλαγές αργότερα όσον αφορά το ύψος του φόρου όσον αφορά τις συναλλαγές συναλλάγματος σποτ. Πολλοί συνάδελφοι πρότειναν να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας. Επί της αρχής συμφωνώ, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μόνο που πρέπει να έχουμε κατά είναι πως η νομική υπηρεσία της ε, Κομισιόν ε, έχει δώσει εδώ πέρα αρνητική γνωμοδότηση ως προς αυτό, λέγοντας πως ε, αντιβαίνει στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Πιθανότατα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια επίσημη γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Όσον αφορά τον καθορισμό του φορολογητέου ποσού στην περίπτωση παραγόγων, μία τροπολογία που πρότεινε ο Πασκάλ. Θεωρώ πως η ιδέα ρύθμισης της ε, φορολογικής βάσης για συμβόλαια παραγόγων έτσι ώστε να φτάσει τουλάχιστον το ύψος μιας άμεσης επένδυσης ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Ταυτόχρονα θεωρώ πως ε, πρέπει να το δούμε το ζήτημα περισσότερο για να είμαστε σίγουροι πως ε, υπάρχουν αρκετές ε, δυνατότητες να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στην πράξη και πως ε, δεν θα οδηγήσει σε υπερβολικές περιπλοκές στον τομέα της εφαρμογής. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω για κάποιες άλλες τροπολογίες. Η ιδέα ιδέα χαμηλότερου ύψους του φόρου για ό,τι γίνεται σε κάποιες ε, πιο διάφανες ε, αγορές, ε, δηλαδή τροπολογία κάρας πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τα ζητήματα έκδοσης και ιδιοκτησίας έχουμε από τους συναδελφούς Κλούπερ, Πέρες, Κανφέν και άλλους αρκετές ε, τροπολογίες για να προσθεθεί η αρχή αυτή της έκδοσης. Θεωρώ επίσης πως καλύτερο είναι να πούμε πως η έκδοση και η αρχή της ε, κατοικίας συμπληρώνουν η μία την άλλη και καλό θα ήταν να μην πούμε ποια από τις δύο υπερισχύει και να δώσουμε και στις δύο ίση αξία για να έχουμε την απαιτούμενη ευελιξία. Τώρα όσον αφορά τις ε, τροπολογίες για ακυρωμένες εντολές ε, της Προέδρου ε, και Πασκάλ Καμφά, τη καλωσορίζω επί της αρχής. Δεν νομίζω πως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει στην πρόταση αυτή, μια που υπάρχουν άλλα αριθμιστικά μέτρα κατά των υπερβολικών ακυρώσεων, αλλά νομίζω πως είναι καλή ιδέα, πρέπει να την εξετάσουμε. Όσον αφορά ένα αποτέλεσμα ντόμινο, της ε, σχεπαπιετικά είναι η τροπολογία, είναι προσωστή κατεύθυνση και το καλωσορίζω και μετά οι τροπολογίες 149 και 50 της κυρίας Πιετικά είναι για την καταγραφή σφαιρολογικές αρχές επίσης ε, της καλωσορίζω, όπως και τις 151, 52, 53 της Sharon Bowles και του Όλε Σμιτ. Νομίζω πως είναι ενδιαφέρουσες και αξίζει να συζητηθούν. Για τους κοινού κανόνες για να μην υπάρξει φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, συμφωνώ πλήρως. Θεωρώ πως οι τροπολογίες αυτές ε, και πάλι είναι ε, και Μπόουλς ε, και Σμιτ μπορούν να γίνουν συμβαστικές τροπολογίες. Η Eurostat ευπρόσδεκτη από εμένα. Όπως επίσης και η διεθνής συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα. Τέλος, μια παρατήρηση για την τροπολογία Giggold για κανόνες περί μη κατάχρησης είναι πάρα πολύ σημαντική, συμφωνώ και τέλος διαχείριση των εσόδων. Θέλω να επαναλάβω πως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζει η πρόταση της Κομισιόν, αλλά θεωρώ ταυτόχρονα πως δεν μπορούμε στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο γενικώ να αγνοήσουμε τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής e ε, να ενισχυθούν οι ήδη πόροι της ε, Ένωσης. Όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, μέρος των εσόδων αυτού του φόρου και όπως και του αναθεωρημένου ΦΠΑ θα πρέπει και θα μπορούσε να πάει στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Θεωρώ πως αυτή η προσέγγιση ε, πρέπει να ενθαρρυνθεί για να εκφράσουμε τη στήριξή μας ε, στο σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το οποίο συνδέεται με τη στήριξή μας στην κοινοτική μέθοδο και θεωρώ πως υπάρχουν πολλές δυνατότητες να επιτύχουμε έναν καλό συνδυασμό και στις αιτιολογικές σκέψεις. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Πρόεδρος, ε, λοιπόν, όταν έχουμε σημαντικά θέματα θα έχουμε και πιο μεγάλο χρόνο ε, ομιλίας ε, για τους σκιώδεις κλπ. Ε, λοιπόν, για να τελειώσουμε στην ώρα μας, ελπίζω ότι οι σκιώδεις δεν θα ξεπεράσουν τα τρία λεπτά στις παρατηρήσεις τους. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά προσπαθήστε. 20 λεπτά πήρε η παρουσίαση της εισηγήτριας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν πάρα πολύ χρόνο οι άλλοι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, μεθοδολογία εργασίας που ακολούθησε, που ήταν πολύ αποτελεσματική και πολύ ε, επαγγελματική. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία. Τώρα, ο πρώτον, όσον αφορά το εναλλακτικό μοντέλο, θα ήθελα να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω για μια ακόμα φορά το γεγονός ε, ότι ο σχεδιασμός ε, του, του, του φόρου αυτού είναι πάρα πολύ ε, σημαντικός γιατί βεβαίως θηλαστικά μπορεί να είναι και η Αγελάδα και το άλογο αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται με διαφορετικό, διαφορετική δουλειά κάνει το κάθε ζώο, άλλου είδους γάλα δίνει το κάθε ζώο κτλ. Ε, και επομένως ε, ε, αυτό ισχύει και για την συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε αυτό το φύχη σίγμα ή αν θα πρέπει να έχουμε ένα τέλος χαρτοσύμου. Όσον αφορά τώρα την, το, το μοντέλο αυτό του, του φόρου πιστεύω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε έτσι ώστε να μην αφήνει καθόλου περιθώρια για φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Ε, όπως ε, αναφέρθηκε και προηγουμένως ε, θα πρέπει να είναι σαφής η αναφορά στην ενισχυμένη συνεργασία. Βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτό το μοντέλο φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και να βασιστούμε και σε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ε, και θα μπορούσε ενδεχομένως να βρεθεί λύση σε πιο προβλήματα μέσα από ε, καλύτερη και μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών. Εγώ είμαι υπέρ ε, του να ε, χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί ο φόρος αυτός ε, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πόροι της κοινότητας. Όμως δεν συμφωνώ με earmarking αυτής της, του φόρου για συγκεκριμένους στόχους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν βεβαίως για ένα σωρό στόχους. Από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρησιμοποιηθούν ε, για ένα σωρό ε, δράσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε για τα δύσκολα θέματα και ε, η συγγήτρια έχει δείξει ήδη καλή διάθεση. Τα δύσκολα σημεία είναι ακόμα ο αποκλεισμός καθώς επίσης και τα συλλεξιωτικά ταμεία ελάχιστη εναρμόνιση ε, και βασιζόμενη και στην ε, ε, πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι μια καλή αρχή. Οι χρηματιστηρικές συναλλαγές είναι επίσης μια καλή αρχή. Και νομίζω ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα, το σημαντικότερο είναι να δούμε, να, να φανεί, μάλλον να διαφανεί ότι έχουμε μια κοινή θέση και ισχυρή θέση και ότι βεβαίως θα θέλουμε ε, να έχουμε και όλη την ε, ε, καλή διάθεση και όλη τη σωστή υποδομή. Τέλος να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια γιατί έχει πάρει κατά την άποψή μας σωστό δρόμο. Είναι καλή η τροχιά την οποία έχει ξεκινήσει και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σάρον. Εξ αρχής να πω ότι η πολιτική μου ομάδα είναι κατά της εισαγωγής αυτού του φόρου. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ κατά, αλλά, αλλά ε, Πρέπει να σας το πω ότι η πολιτική μου ομάδα δεν θα στηρίξει ε, την ε, πρόταση της Επιτροπής. Ε, βεβαίως μπορώ να συμφωνήσω ότι με το, με το γεγονός ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να συμβάλλει με κάποιο τρόπο. Ε, και να αποκαταστήσει τις ε, ζημιές. Τώρα, ε, γιατί θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά εδώ. Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε απλώς ε, θα, δοθούν τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι λένε ότι τα χρήματα ε, θα δοθούν για αναπτυξιακά προγράμματα, για θέματα, για προγράμματα που σχετίζονται με την ε, κλιματική αλλαγή κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να πιστούμε για, τα επιχειρήματα αυτά. Το, το πιο σημαντικό θέμα, σημείο είναι ότι βεβαίως πρέπει να πληρώνεται ένα ένα είδος φόρος ε, και όταν αγοράζει ψωμί πληρώνει ε, ε, ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι εάν εισαχθεί ο φόρος αυτός θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η αρχή του ε, κατοίκου, ε, του resident ε, θα καλύπτεται και στην προκείμενη περίπτωση. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε σε περίπτωση των διεθνών συναλλαγών εάν υπάρχει ας πούμε στη Βραζιλία μία, μία συναλλαγή στην οποία εμπλέκεται και κάποιος Ευρωπαίος εταίρος θα πληρωθεί ο φόρος ή όχι το σημαντικό είναι γενικά να δούμε ε, εάν θα μπορέσουμε να ε, διαχειριστούμε τον όγκο των συναλλαγών γιατί είναι εκατομμύρια οι συναλλαγές και γίνονται ταυτόχρονα. Υπάρχει ε, ασφάλεια όσον αφορά τη δυνατότητα αντιμετώπισης διαχείρισης των συναλλαγών αυτών και αν ε, κάτι τέτοιο είναι σημαντικό θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί ίδιο, ε, ίδιο, ε, ίδιο τόκος, ίδιο ποσοστό της 100 για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωπικά μπορώ να στηρίξω τους στόχους, τουλάχιστον θεωρητικά πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, αλλά πρακτικά υπάρχουν ακόμα πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αποσαφινιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας εξοικονομήσω λίγο χρόνο. Γιατί είμαι μεταξύ αυτών που κατέθεσαν τροπολογία, μια τροπολογία για την απόρριψη της θέσης της Κομισιόν. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα. Καταλαβαίνω ότι σήμερα συζητούμε τροπολογίες, όχι βασική συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του σχεδίου αυτού. Εμείς λοιπόν είμαστε κατά και θα παραμείνουμε υπέρ της απόρριψης. Ακούγοντας την κυρία Ποδηματά, εκτιμώ την, το έργο της και τις εξηγήσεις της, αλλά ακόμα και μετά από αυτά που είπε, εξακολουθούμε να θέλουμε να απορρίψουμε. Ο Πασκάλ. Ναι, για τα κύρια σημεία τα οποία αναφέρθηκαν στη συζήτηση <clears throat> για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Άννη, είναι θέμα υποδείγματος. Πρέπει να φορολογήσουμε τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές και αυτό που θέλουμε από τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι να είναι μακροχρόνιοι επενδυτές είναι σε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μοντέλο, αυτό δεν θα οδηγήσει σε προβλήματα τα συντοξιδευτικά ταμεία. Για ένα ταμείο σε σχέση με την προσθέμενη αξία. Και αυτό αναφέρθηκε στο, στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο φόρος δραστηριοτήτων λοιπόν είναι ένα διαφορετικό μοντέλο. Και το πρόβλημα με το φόρο αυτό είναι ότι, είναι ότι τα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, τις συναλλαγές οι οποίες έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα για την πραγματική οικονομία. Ενώ ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών διαφορίζει μεταξύ αυτών που είναι πάρα πολύ βραχυπρόθεσμες και κερδοσκοπικές από αυτές που εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία. Επομένως δεν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με το φόρο δραστηριοτήτων και δεν επιτυχάνουμε τον ίδιο στόχο. Δεν είναι λοιπόν δύο πράγματα τα οποία είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους. Για την επιλογή τώρα που έκανε η Κομισιόν για τις ε, αλλαγές, ε, για τις ε, αγορές κεφαλαίου η Κομισιόν έχει πει ότι αυτό είναι κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Θα ήθελα όμως να έχω και μια μελέτη που δείχνει πώς καταλήγει η Κομισιόν σε αυτό το συμπέρασμα ότι ξεφεύγει από τις ε, δυνατότητες συνθήκες, γιατί είχαμε στο παρελθόν μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πριν από μερικά χρόνια που έλεγε το αντίθετο. Εγώ δεν είμαι νομομαθής, δεν έχω καταρχήν μια άποψη στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να δω όμως και ποια είναι η επιχειρηματολογία της Κομισιόν, η οποία δικαιολογεί μια εξαίρεση των αγορών συναλλάγματος. Περιμένουμε επίσης και τη μελέτη αντικτύπου για την οικονομική ε, ανάπτυξη από τον Επίτροπο ο οποίο είναι αρμόδιος για τα θέματα φορολογίας. Θα, ήθελα... θα θέλαμε η Κομισιόν το να μα δώσει στοιχεία για αυτό και για να απαντήσω σε αυτά που ανέφερε ο Βολφ Κλίντς με ποιο τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αρχή της ε, εντοπιότητας του κατοίκου ότι κάποιος είναι πραγματική εκεί θα πρέπει να προσθέσουμε και την αρχή της μεταβίβασης μιας ιδιοκτησίας. Αν κάνετε λοιπόν μία συναλλαγή στην Σιγκαπούρη και δεν τη δηλώνετε, για να μην πληρώσετε φόρο, τότε ο τίτλος αυτός που αγοράζετε δεν είναι έγκυρος και παίρνετε ένα νομικό κίνδυνο που καμία τράπεζα δεν θέλει να τον αναλάβει. Έτσι, προσθέτοντας την αρχή της ιδιοκτησίας η οποία κτείται, τότε μπορούμε να ενισχύσουμε την αρχή του κατοίκου. Οι συναλλαγές τώρα γίνονται με εντολές, γίνονται όλα αυτά σε καταχωρη, καταχωρημένες σε αγορές, δεν είναι στην αγορά, σε εκτό, δεν εκτός αγοράς, ε, εκτός οργανωμένων αγορών και μπορούμε για τις ε, ε, συναλλαγές που γίνονται με μεγάλη ταχύτητα και συχνότητα να δούμε ποιες από τις εντολές που βρίσκονται σε ένα καρνέ εντολών έχουν πληρωθεί ή όχι και με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να ξέρει ποιες είναι αυτές οι οποίες έχουν εκτελεστεί και ποιες όχι, επομένως ποιες από αυτές θα πρέπει να υπόκεινται σε φορολογία. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε και μία διαφάνεια. Ό,τι καταγράφεται λοιπόν σε οργανωμένε αγορέ δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα για την εφαρμογή αυτού του φόρου. Ο Μίγελ Πόρτους. Πιστεύω ότι η συγγήτρια όταν έλαβε το λόγο σε μια συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές είπε κάτι πολύ σωστό, ότι μέχρι τώρα η δραστηριότητα της Επιτροπής μας είχε σαν στόχο να εξασφαλίσει την ε, εμπιστοσύνη της αγοράς. Για πρώτη φορά αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για το πώς θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ακριβώς αυτό θα πρέπει να είναι η κύρια πολιτική γραμμή, ο κύριος πολιτικός άξονας της προσπάθειάς μας σε αυτό το θέμα, για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και γι' αυτό το λόγο, παρά το γεγονό ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν για ένα νέο κανονισμό, εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε και κάποια αναφορά στην ιδέα ότι αυτός ο φόρος θα πρέπει να εισπράτεται σε εθνικό επίπεδο μεν, αλλά θα πρέπει να καταστεί ένας πόρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού και να χρησιμοποιείται για πολιτικές οι οποίες αντιμετωπίζουν την ένδια την κλιματική αλλαγή και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Τούτου λεχθέντος, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα νέο εργαλείο το οποίο θα πρέπει να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα ε, και μεταφέρει πόρους από το κεφάλαιο στην εργασία. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι εγώ δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι πρώτα του να έχουμε δύο φόρους που έχει παρουσιαστεί από την Κομισιόν επιτυγχάνει τους στόχους τους οποίους επιδιώκουμε, δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση των επενδύσεων την ανακατεύθυνση των επενδύσεων. Πιστεύω. Υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και οι οποίες και αυτές θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας. Και το 0,001% είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό επίσης κατά την απόψη μου αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνω. Μια τρίτη παρατήρηση, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Πασκάλ Καμφέαν προηγουμένως. για την ανάγκη να εδρεωθεί η αρχή της, του κατοίκου με την αρχή της ιδιοκτησίας που αποκτάται από ένα τίτλο και επίσης συμφωνώ με αυτά που λέει η συγγήτρια σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Πιστεύω ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να δώσει κίνητρα σε μια πιο συντηρητική συμπεριφορά από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και όχι μια επιζήτηση κινδύνων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν πρόκειται για συνταξιδοτικά ταμεία. Τρία λεπτά μου μίλησα να, μου ζητήσετε να μιλήσω, τρία μίλησα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Η Αστρίδ Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι πεπισμένη για τα λεγόμενα καλά αποτελέσματα που θα μας φέρει ε, αυτή η φορολογία, αλλά έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες ε, έτσι ώστε ε, τα OPSVM των συνταξιδοτικών ταμείων που ανταποκρίνονται σε κριτήρια υπάρχουσας οδηγίας να εξαιρεθούν, λέω. Ε, λυπούμε που δεν θέλει να το δεχτεί αυτό η, ε, συγγήτρια γιατί είναι ένα μέτρο πολύ λογικό, απλής λογικής ε, γιατί αναφέρεται σε ε, μέσα τα οποία ε, είναι μέσα αποταμίευσης τα οποία χρησιμοποιούν ε, πάρα πολύ ε, και που βεβαίως αφορούν κάποια αποταμίευση μακροπρόθεσμη με τελικό σκοπό και την κοινωνική προστασία. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, αλλά δεν είναι δυνατόν να τιμωρούνται επενδυτικά ταμεία τα οποία εκ της τους καλούνται να τζιράρουν το, το, ταμείο τους αυτό ε, και για κάθε κίνηση να πρέπει να πληρώνουν αυτό το φόρο. Επίσης, ε, ε, για πολλές περιπτώσεις, σαν αυτές που ανέφερα προηγουμένως αλλά και άλλες, θα μπορούσε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα ντόμινο το οποίο θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μπορούσε να έχει μεγάλη επίπτωση σε, όλες τις, σε όλο το επενδυτικό τοπίο ε, και βεβαίως ε, θα στραγγάλιζε και τους επενδυτές και τις τράπεζες απέναντι σε ε, ξένους άλλους επενδυτές που δρούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εάν κατάλαβα καλά αυτά που είπε η συγγήτρια, ε, φαίνεται ότι αμφισβητείται κατά κάποιο τρόπο και μια γερμανική μελέτη η οποία λέει ότι ε, εάν για 40 χρόνια κάθε φορά επένδυε κάποιος 100 ε, ευρώ τελικά θα είχε μία μείωση στο τέλος της περίοδου, της περίοδου αυτής 14.000 ευρώ. Ε, εάν βεβαίως εφαρμοστεί ε, και σε αυτές τις συναλλαγές επενδύσεων σε κινητές αξίες ή ε, θα μπορούσε να έχει αυτήν την επίπτωση και εν πάση περιπτώσει εάν πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ο στόχος αυτός τουλάχιστον θα πρέπει να ληφθεί δράση κατά αυτών των στρεβλωτικών και πιο ανησυχητικών ας πούμε φαινομένων. Η... επίσης πρέπει να πω ότι και οι συγγήτρια και οι συνάδελφοι που τη στηρίζουν φαίνεται ότι βρίσκονται σε μια διαφορά φάσης σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο Συμβούλιο και ο κύριος Σόιμπλε, επικεφαλής πολλών ε, άλλων, κατέδειξε και είπε σαφώς ότι ε, έχει ξεχαστεί, έχει θαυτεί αυτή ε, η διαδικασία φορολόγησης. Ίσως θα πρέπει να προσπαθούμε λίγο ε, να μην μας ξεπερνούν τα γεγονότα και να μην είμαστε διαφοραφάσεις με την πραγματικότητα. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω το ίδιο πρόβλημα όπως ο κύριος Κλίντς προηγουμένως. Εγώ έχω την άποψη που έχει το δικό μου Εθνικό Πολιτικό Κόμμα. αν αφήσουμε τις ε, <clears throat> τροπολογίες απόρριψης. Βλέπετε ότι πολλοί από εμά θέλουν να υπάρξει κάποια μορφή φορολογίας για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτοί που απορρίπτουν τη συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν την απορρίπτουν γιατί τη θεωρούν μη επικοδομητική. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να, έχουμε, να είχαμε και μια συζήτηση του τι θα γινόταν αν αυτό το σύστημα την χανε απόρριψης. Αλλιώς θα πάψουμε να έχουμε κάποιο λόγο σε σχέση με αυτά τα οποία θα γίνουν στη συνέχεια. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την εισηγήτρια και επίσης από την πρόεδρό μας το εξής. <clears throat> Επειδή εμεί υποτίθεται ότι θα ψηφίσουμε στις 25-26 Απριλίου, στο τέλος Απριλίου, είναι σόφρον αυτό, μήπως θα πρέπει να περιμένουμε λίγο περισσότερο. Πάντα προσπαθούμε να έχουμε παραλληλισμό στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι αυτή την Παρασκευή στην συνεδρία του Συμβουλίου στην Κοπεχάγη θα προκύψουν και κάποιες αλλαγές στην πρόταση Κομισιόν. Μήπως θέλετε να έχετε κάποια θέση αναδίπλωσης, ρωτάω την εισηγήτρια. Αυτό είναι πάντα χρήσιμο. Δεν θα σταθώ τώρα στα επιχειρήματα γιατί όπως σας είπα δεν είμαι κατά των φόρων, αλλά είμαι ε, εναντίον φόρων που δεν θα αποδειχθούν θετικοί στην πράξη. Και πρέπει να έχουμε μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Και αυτό είναι και ένα ερώτημα για τον κύριο Κλίνς, ο οποίος έχει φύγει. Πώς θα συμμετάσχουν οι Ευρωζώνοι, λιγότεροι, Λιγότερε χώρε από τα μέλη της Ευρωζώνης. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσοι θα συμμετέχουν σε αυτό το φόρο και δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Η ΚΕΙ, e ναι, πάρα πολύ. Σύντομα. Δεν θα παρέμβαινα, αλλά ε, ακούγοντας αυτό το θέμα για το τι, για την εξαίρεση των συνταξιοδοτικών ταμείων, η συγγήτρια Άννη, Άννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν ένα άτομο που έχει διαχειριστεί συνταξιδοτικά ταμεία, όσο πιο, όσο πιο συντηρητικό είναι ένα ταμείο, τόσο πιο συντηρητική είναι η επένδυσή του, θα πρέπει να κάνει και αντισταθμίσεις, hedges, δηλαδή θα πρέπει κάθε μέρα να κάνει κανείς εκατοντάδες συναλλαγές για να έχει την αντιστάθμιση κινδύνου. Αν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα μπορεί, αν ο φόρος εφαρμοστεί δεν θα μπορεί ένα χαρτοφυλάκιο να παραμένει συντηρητικό. Αν γίνει πιο επικίνδυνο το χαρτοφυλάκιο με εισαγωγικά γιατί κοστίζει πολύ η αντιστάθμιση, τότε αυτό θα επιβαρύνει πολύ περισσότερο το συνταξιοδοτικό ταμείο. Και η έρευνα αυτή τη Γερμανία έδειξε ότι θα είναι τεράστια η επιβάρυνση για ένα συνταξιοδοτικό ταμείο. Επίση στη Σουηδία και στην Ολλανδία μελέτε έδειξαν ότι σε μια επένδυση 20 ετών θα υπάρξει επιβάρυνση 20%. Αν σκεφτείτε ποιο είναι το κόστος για κάθε εταιρεία που θα πρέπει να πληρώσει αυτό το φόρο για αντιστάθμιση κινδύνου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιό του. Μπορεί να χρειάζεται για κάθε συναλλαγή να πληρώνει κανείς 20, μέχρι 27 φορές το φόρο γιατί κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή απαιτεί μια πλειάδα συναλλαγών αντιστάθμισης. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα. Όσο συντηρητικό είναι ένα χαρτοφυλάκιο, τόσο πιο πολύ θα κοστίσει. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καταλάβετε ότι έτσι δουλεύει η διαδικασία δυναμική αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια. Σβέν. Όχι, δεν θέλει, λέω Σβέν. Θα έλεγα το ίδιο που έλεγε η Κέι. Σε πολλές περιπτώσεις οι κανονισμοί μας μας υποχρεώνει να κάνουμε αντιστάθμιση κινδύνου. Γιατί αλλιώς παίρνουν υψηλότερη στάθμιση κινδύνου και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν περισσότερα κεφαλαιοχικά αποθέματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μας σκεφτείτε το Solvency 2 και το ρόλο των συνταξιοδοτικών ταμείων. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν δεν θέλει κανείς να εξαιρέσει γενικά τα συνταξιοδοτικά ταμεία, ίσως θα πρέπει να σκεφτεί κανείς για το πώς θα πρέπει να εξαιρείται η απαραίτητη αντιστάθμιση κινδύνου που ήταν αυτό ακριβώς που προτείναμε για ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάποιες θεσμικές ανάγκες αντιστάθμισης κινδύνου και επομένως θα έδινα και στα συνταξιδοτικά ταμεία το ίδιο επίπεδο προστασίας. Γιατί αλλιώς ε, περιορίζει κανείς τις μακροχρόνιες επενθύσεις και την ανάκαμψη. Δεν θέλουμε μία, αν δεν θέλει κανείς μία συνολική ε, εξαίρεση, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο μιας πιο συγκεκριμένης εξαίρεσης για να λυθεί το πρόβλημα των επενδύσεων. Γιατί δεν, η αντιστάθμιση κινδύνου δεν είναι κερδοσκοπία. Πολλές φορές είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς και στην πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Σέμετα δεν ήξερε ο Επίτροπος ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία κάνουν τέτοιες αντισταθμίσεις και δεν ξέρω αν και η Γενική Διεύθυνση φορολογία το καταλαβαίνει αυτό και πρέπει να μιλήσει με την Γενική Διεύθυνση για την αγορά. Αλλιώς θα πρέπει στους κανονισμούς μας να σταματήσουμε να ζητάμε αντιστάθμιση κινδύνου και να ζητήσουμε από τους διαχειριστές των ταμείων να χρησιμοποιούν το νιονιό τους, κάτι το οποίο εγώ θα το υποστήριζα. Αλλά πολλοί νομίζω ότι θα νιώθανε πανικό αν γινόταν κάτι τέτοιο και έπαβε να υπάρχει αυτή η ανάγκη αντιστάθμισης κινδύνου. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω ήταν η, η έννοια της κοινή ευθύνη. Αλέγγυας ευθύνη σίγουρα. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν καλό να υπάρχει η ανάγκη να, έχει, να φέρει κανείς ευθύνη για πράξεις που έκανε ένας επενδυτής ή μια τράπεζα που δεν πλήρωσε τους φόρους. Δεν μπορεί ένας συναλλασσόμενος να φέρει ευθύνη για τις πράξεις του, ε, του άλλου συναλλασσόμενου και να, να θεωρηθεί ότι, είναι, ότι έχει αστική ευθύνη. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε καταχρήσεις εξάλλου. Και αυτό αναφέρεται και σε κάποιες τροπολογίες που έχω καταθέσει. Αν δεν υπάρχει τώρα κάποιος άλλος που θέλει να λάβει το λόγο, Άννη, έχεις ακόμα δύο λεφτά με την ανοχή και των διερμηνέων. Yes, uh, it will be just for two minutes, just to thank you all for... Δύο λεπτά μόνο. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια. Βλέπω βέβαια ότι πολλοί από τους ε, ε, σκιώδεις έχουν ήδη εγκαταλείψει την αίθουσα, δεν πειράζει. Όπως είπα και στα αρχικά μου σχόλια, Ε, συζητούμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες όσον αφορά τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όσον αφορά μια σφαιρική συμφωνία. Την ιδέα επίσης ε, της χρήσης των εσόδων, όσον αφορά ένα ζήτημα το οποίο εστιάζει, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησής μας, είναι αυτό το οποίο αφορά τις ε, προτάσεις εξαίρεσης των συγκριτικών ταμείων. Εγώ νομίζω ότι ήμουν απολύτως ακριβής και επεξήγησα πολύ τη θέση μου ε, βάσει μελετών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ξέρω ότι θα υπάρχουν βέβαια και κάποια πιο καινούργια στοιχεία κατά αυτήν την έννοια. Ένα τελικό στοιχείο. Με προβληματίζει, με προβληματίζει λέω, γιατί όλες αυτές οι ανησυχίες που αναφέρθηκαν εδώ σχετικά με τα συνταξιδετικά ταμεία και ζητούν ε, να μην εγγραφεί στο πεδίο της ε, οδηγίας ε, το θέμα των συνταξιδετικών ταμείων, ε, τελικά αντιτίθενται πλήρως τα σχόλια αυτά στα όσα αναφέρονται στο προήμιο ε, του, της οδηγίας για, το, το, για τον φόρο χρηματοδοτήσεων το πιστοτικών συναλλαγών. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά την προσέγγιση αυτή. Νομίζω ότι όσον αφορά τις διαφορετικές ευαισθησίες ε, ε, σχετικά με τα χρήματα τα οποία ε, αποταμιεύουν οι συνταξιούχοι στα συνταξιωτικά ταμεία, προφανώς δεν αποτελούν προνόμιο μερικών. Όλοι μας ανησυχούν. Σχετικά με το ερώτημά σου να σου πω ότι ε, μερικοί μου είπαν σταμάτησέ το γιατί θα λειτουργήσει στο τέλος. και πιστεύω ότι τελικά εάν ε, όπως οι περισσότεροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν ε, εάν πραγματικά υπάρξει αυτός ο φόρος συναλλαγών ε, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν και κάποια αντισταθμιστικά μέτρα έτσι ώστε να μετριαστεί η επίπτωση που μπορεί να έχει σε ορισμένε κατηγορίες πολιτών. Λοιπόν, θα συζητηθεί πάντως το θέμα αυτό τον, την επόμενη εβδομάδα στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ και ενδεχομένως θα έχουμε και κάποια νέα στοιχεία όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου, τη στάση μάλλον του Συμβουλίου. Και διαφορετικά η 25η Απριλίου, όπως μας είπε και η συγγήτρια, θα είναι ο, ο χρονικός μας στόχος. Λοιπόν, αυτή δεν είναι διαδικασία συναπόφασης. Και επομένως δεν έχει και πολλή έννοια να αναβάλουμε την ε, συζήτηση έτσι ώστε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα του Συμβολίου. Αντιθέτως πιστεύω ότι καλύτερο θα ήταν να έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψή μας ως, ε, ως σώμα όσο γίνεται πιο έγκαιρα και πιο ε, Πολύ ωραία. Και όσον αφορά την Ολομέλεια, ε, έχουμε στόχο τη 2 του Μαΐου ή την 1 του Ιουνίου. Αυτά ε, για σήμερα θα τα πούμε αύριο. Okay, 9 o'clock tomorrow morning. And also, and also yes, and coordinators as well.